εμείς όμως να μας βλέπουν με καλό μάτι. πολλές εφημερίδες γράφουν κακά πράγματα για μας και πολλοί κόσμος αναρωτιέται μα τι στο καλό χρειάζονται όλοι αυτοί στην Ευρώπη. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που είμαστε εδώ για να εργαστούμε, για να αποδείξουμε ότι σε κάτι είμαστε χρήσιμοι. Όσον αφορά στις ανακοινώσεις του Προέδρου, μία και μόνη ανακοίνωση σημαντική για τους συντονιστές. Υπήρξε, υπήρχε μία ερώτηση για, ε, της Επιτροπής για την εκτόξευση του δορυφόρου και μας είχαν καλέσει να πάμε στο Κουρού. Είχαμε δεχτεί την πρόσκληση η διάσκεψη των Προέδρων είπε ναι αλλά μόνο ένας βουλευτής να πάει. Πολύ καλά, μας δόθηκε η άδεια. Θα ήθελα να γραφτεί στα πρακτικά ότι η διάσκεψη των προέδρων είναι αυτή που αποφάσισε πόσα άτομα μπορούν να πάνε. Δηλαδή υπήρξε ανάμειξη της ε, Τη διάσκεψης των Προέδρων για το πώς εμείς ελέγχουμε τον προϋπολογισμό μας. Δεν θέλω να ξεκινήσω κανέναν καυγά βέβαια, το ετονίζω όμως και πρέπει να αποφασίσουμε για το ποιος θα πάει. Θα πρέπει να το συζητήσουμε και στα πλαίσια των ομάδων σας για να δούμε ποιον θα στείλουμε. και όποιος είναι να πάει να ε, κλείσει και τη το αεροπλάνο του και να μην αφήσει να σέρνεται η υπόθεση. Τώρα για τα πρακτικά όμω και για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα θα πρέπει να πούμε ότι δεν δεχόμαστε να ορίζει κάποιο άλλο το πώ θα καθορίσουμε τον, προσ... τον προπολογισμό μα, την κατανομή του προπολογισμού μα. Τώρα λοιπόν έχουμε τι οδηγίες με τα σχετικά νούμερα στα έγγραφά μα. Θα τι συζητήσουμε όχι μόνο γενικά αλλά και πιο ε, εξειδικευμένα και στη συνέχεια θα δούμε θα δούμε εάν αυτές οι περιπτώσεις έχουν συνέπεια στην η υπόθεση αυτή και αν μπορούν να αποτελέσουν μια κατάλληλη βάση για την υπόθεση. Πρέπει να κάνουμε ανάλυση δηλαδή για να δούμε αν είναι μια σωστή επιλογή ή όχι. Και γι' αυτό θα ήθελα και να εκφράσω ε, την ικανοποίησή μου για το ότι ο Πολ Χάτσον από τη Γενική Διεύθυνση της Ενέργειας είναι παρόν εδώ για να μας δώσει μια πρώτη εικόνα αυτής της αξιολόγησης θα δώσω ένα στον Κλωτ Τούρμες ως, προ, εισηγητή πρώτο το λόγο και στη συνέχεια θα δούμε και τις απόψεις σας και τις ερωτήσεις σας. Έχουμε περιθώριο, έχουμε χρόνο. Είναι θα μπορούσαμε να έχουμε ακυρώσει κιόλα τη συνεδρίαση, να την έχουμε περικόψει, αλλά πάντως ήταν καλή ευκαιρία πιστεύω να ε, δούμε, αφού έχουμε αρκετό χρόνο, το θέμα στις λεπτομέρειες του. Κύριε Χάτσον, εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλημέρα. Θα πω δύο λόγια για την πρόταση για να εξηγήσω μετά την ε, αξιολόγηση επιπτώσεων. Συμμεριζόμαστε την άποψη του κύριου Ρόιλ ότι είναι σημαντικό αυτή τη χρονική στιγμή να εξασφαλίσουμε την στήριξη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και ένα τρόπος να το καταφέρουμε αυτό είναι να βοηθήσουμε τον πολίτη να μειώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Αυτό νομίζω θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη αν το καταφέρουμε. Βέβαια, ο κύριος στόχος είναι η, ε, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περικοπή κατά 20% ε, των δαπανών σε ενέργεια, της ε, δαπάνης ενέργειας μέχρι το 2020 που όπως φαίνεται ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί. Μέχρι 10% περικοπή μπορούμε να καταφέρουμε ε, με την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Συζητήσεις υπάρχουν ακόμη σε επίπεδο και συμβουλίου. Τίθεται και το ζήτημα αν θα πρέπει να υπάρχουν εθνικά δεσμευτικοί στόχοι. Προσέγγιση την οποία είχε ε, ακολουθήσει και η έκθεση του κυρίου Μπένσον που ήθελε το κοινοβούλιο πέρυσι. Αλλά το Συμβούλιο δεν ακολούθησε την ίδια ε, επιλογή. Στο σχέδιο οδηγίας που έχετε ενώπιόν σας έχουμε μια προσέγγιση σε δύο στάδια η πρόταση δηλαδή περιλαμβάνει μια σειρά δεσμευτικών μέτρων, όχι στόχων, μέτρων δεσμευτικών, που κρίνουμε και με βάση και τη μελέτη αξιολόγησης ότι θα μας επαναφέρουν στην τροχιά του στόχου 2020 και 20%. Εάν όμως μέχρι τις αρχές του 2014 δεν έχουμε προχωρήσει όπως προβλέπετε, τότε επανέρχεται η Επιτροπή με μια πρόταση για δεσμευτικούς πλέον στόχους. Ποια είναι τα δεσμευτικά μέτρα. καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας. Έχουμε προτάσεις και για τον ε, δημόσιο τομέα. Μπορεί και αυτός να δραματίσει ένα ρόλο ηγετικό ως προς την, ε, ως προς την ε, αγορά επαραδείγματη της δημόσιας προμήθειας μόνο αποτελεσματικών ως προς τη χρήση ενέργειας ακινήτων ή εξοπλισμού και βέβαια με την ανακαίνιση των κτηρίων του Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο συγκεκριμένο εξοικονόμησης ενέργειας από τους πελάτες ή τα κράτη-μέλη θα πρέπει τα ίδια να βρουν ένα διαφορετικό τρόπο για να εξοικονομήσουν τον πόρο αυτόν, τον, το ποσοστό αυτόν. Στο άρθρο 8 εξασφαλίζεται καλύτερη ενημέρωση για τον μικρό καταναλωτή, τον ιδιώτη καταναλωτή ως προς την ε, ε, τις λεπτομέρειες του λογαριασμού του, του ηλεκτρικού, στο άρθρο 10, έχουμε περισσότερη αξιοποίηση, αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας και μετά έχουμε στο 12 την διαχείριση των δικτύων. Νομίζω ότι με αυτά, γιατί υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, με αυτά μπορώ να σας δώσω μια γενική εικόνα των προθέσεών μας. Τώρα, τι, δίνουν, ε, τι μας δίνει η μελέτη επιπτώσεων ως προς τις προτάσεις αυτές. Καταρχάς, η μελέτη επιπτώσεων επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι δεν θα πετύχουμε το στόχο όπως πάμε. Και ότι θα ε, έχουμε φτάσει το 2020 σε 1942 ε, όγκους ε, πετρελαίου ενώ θα έπρεπε να είμαστε στο 1500 περίπου ή κάτω από το 1500 μέχρι το 2020. Αυτό με βάση και τα έγγραφα που ε, στηρίζουν τη μελέτη. Δεύτερον, δεν έχουμε μόνο τις ε, επιλογές πολιτικής που σας έχω περιγράψει, αλλά και άλλες επιλογές πολιτικών αποφάσεων ή αντιδράσεων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση ε, σε σχέση με το πρόβλημα και την ανάκτηση του στόχου για το 2020. Δεν έχω αρκετό χρόνο για να σας δώσω τις εξηγήσεις του κάθε ενός από τα μέτρα αυτά ή τις επιλογές αυτές, αλλά μέσα στο έγγραφο υπάρχουν στην μελέτη αξιολόγηση. Τρίτον, και εδώ δεν θα πρόκειται εξάπαντος να σας δώσω τις λεπτομέρειες αυτού του πίνακα, έχουμε μια ολόκληρη ε, σειρά πιθανών συνεπειών καταγράψει με διαφορετικά μοντέλα το μοντέλο Prime και το EFME e, που γνωρίζετε φαντάζομαι και με ένα τρίτο μοντέλο, το BIM λεγόμενο μοντέλο ακτίνα που μας επιτρέπουν να καταγράψουμε συνέπειες και επί του ΑΕΠ και επί της κατανάλωσης των επενδύσεων, εισαγωγών, εξαγωγών, τιμών καταναλωτού, εκπομπές αέριων ε, ε θερμοκηπίου, τιμές ως προς τις ανταλλαγές εκπομπών και ούτω καθεξής. Και συνεχίζουμε επί τη βάση αυτής της αξιολόγησης με τον εντοπισμό των στόχων που θεωρούμε ότι θα είναι οι πιο αποτελεσματικοί για των επιλογών καλύτερα, που θα είναι πιο αποτελεσματικές για την επίτευξη του στόχου του 2020. Και προσπαθούμε να διαγνώσουμε το ρόλο που θα έχουν συνολικά σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν δηλαδή την εξέλιξη συνολικά. Φέρει πίν με καλύτερη αποτελεσματικότητα ε, για τα δημόσια κτίρια μπορεί να είναι μέτρα που θα επιτύχουν αυτό, τα οποία θα ταυτίζονται με τα μέτρα για την καλύτερη ε, για την αγορά εξοπλισμού πιο αποτελεσματικού ή πιο οικονομικού σε ενέργεια. Αυτές τις επικαλύψεις τις λαμβάνουμε υπόψη και κοιτάμε εάν όντως τα μέτρα αυτά μπορούν να μας οδηγήσουν στους στόχους που θέλουμε. Βλέπουμε ότι θα μας επιτρέψουν να επανέλθουμε στην στοχοθέτηση του 2020 με ένα ποσοστό σφάλματος ε, μικρό. Επίσης, η εξοικονόμηση ορίζεται ότι θα προέρχεται κατά 40% από την προσφορά και 60% από τη ζήτηση, δηλαδή πιο αποτελεσματική ε, παραγωγή ενέργεια στο 40% και αλλαγή συμπεριφοράς ή πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ενεργειακών μας αναγκών, ικανοποίηση των ενεργειακών μας αναγκών κατά 60%. Και βλέπουμε επί του ΑΕΠ μια ελαφρώς θετική επίπτωση και μια ελαφρώς θετική επίπτωση επί της απασχόλησης. Χρειάζεται φυσικά σε αυτές τις ε, δυσχερείς οικονομικές περιόδους να έχουμε και θετική οικονομική επίπτωση όποιων μέτρων εισάγονται. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σχετικά θετική επίπτωση, περιορισμένη με αλλά θετική. και επίσης ε, μπορεί να υπάρχει μια ε, ασήμαντη μένα αλλά θετική και μια κάποια αναδιανεμητική επίπτωση ως προς το εισόδημα των νοικοκυριών. Βλέπουμε επίσης ως προς την κατανομή αυτών των ε, των ωφελιών ότι γενικά οι τομείς της οικονομίας αποκομίζουν όφελος από την εισαγωγή των μέτρων αυτών και σε μια, σε μια γενική αξιολόγηση όλων των μέτρων Βέβαια, μιλάμε για μέτρα τα οποία για να τα αναπτύξει κανείς πρέπει να καταβάλει το σχετικό κόστος. Ξεκινώντας δηλαδή την εφαρμογή έχουν δαπάνη, αλλά στα 10, 15, 20 χρόνια, ανάλογα με τη διάρκεια του μέτρου που ε, προτείνεται, ε, θα έχουμε θετικές, ε, θετικό αντίκτυπο. Και προχωρώντας, πριν κλείσω αυτή πολύ σύντομη ε, μελέτη, για να σας δώσω μετά και τις ε, απαντήσεις όποιες ερωτήσεις έχετε, πολύ σημαντική πτυχή είναι το να δούμε το πώς αυτή η πρόταση ε, διασυνδέεται με υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και δει με το σχήμα ETS της ανταλλαγής εκπομπών. Είδαμε με διαφορετικά μοντέλα διαφορετικές απαντήσεις ή μάλλον για να ξεκινήσω διαφορετικά και τα δύο μοντέλα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτό το σύνολο πολιτικών μέτρων συμπληρωματικά με τα όσα ήδη ισχύουν οπωσδήποτε θα μας οδηγήσει σε εξοικονόμηση εκπομπών αέριων θερμοκηπίου. Άρα δεν θα αναδιανεμηθεί απλώς ε, ε, ο τομέας των ε, αερίων θερμοκηπίου, δεν πρόκειται απλώς να αλλάξει αναλογίες εσωτερικά μέσα στον τομέα, αλλά θα έχουμε σημαντικές αλλαγές και αντίστοιχα τιμές σημαντικά μειούμενες των ε, ETS, των ε, ανταλλαγών δηλαδή, με βάση το ένα μοντέλο σχεδόν μηδενικές και με βάση το άλλο, το Primes, μικρή μείωση μόνο ως προς το τίμημα του ETS, δηλαδή περί τα 2 ευρώ ανατόνο αλλά πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα είναι τέτοια που δεν μπορεί να καλυφθεί με απλώς ε, διαφορετικές προσωμιώσεις. Άρα πρέπει πολύ προσεκτικά κατά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας να παρακολουθούμε το συγκεκριμένο τομέα. Αυτά, Πρόεδρε. Ε, δεν ήθελα να σας ε, καθυστερήσω περισσότερο. Έχουμε 1.400 σελίδε όμω, υλικό και τεκμηρίωση για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει. Ευχαριστώ, Λέω ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι ούτω ή άλλω είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ξέρουμε ποια είναι η βάση αυτή τη απόφαση. Είναι κάτι το πολύ ευρύ και το πολύ σημαντικό. Α ξεκινήσουμε όμω ε, τώρα με τι παρεμβάσει των συναδέλφων και πρώτο ο κύριο Τουρμέσο ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη είναι εξής. Εάν αντελήφθην σωστά την ε, μελέτη επιπτώσεων, μιλάτε για 200 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. Το άρθρο 6 με την υποχρέωση δηλαδή για τις ε, ενεργειακές επιχειρήσεις και ε, διανομής ενέργειας μιλάει για 100-110 δισεκατομμύρια. Αυτή λοιπόν η συνέπεια η συγκεκριμένη θα είναι το μεγάλο κομμάτι της εξοικονόμησης και μετά θα έχουμε μικρά-μικρά από εδώ και από εκεί. Τα 110 με 20 περίπου αυτά δισεκατομμύρια τόνοι συμπεριλαμβάνονται επίσης στην παράγραφο 6-9 η οποία από ό,τι άκουσα πρωτοεμφανίστηκε από την πρώτη μέρα των ε, συναντήσεων με το opt-out ουσιαστικά και μεταξύ πρώτης ημέρας των συναντήσεων των εκπροσώπων της Επιτροπής και της ημέρας όπου συνεδρίασαν οι σεφ του καμπινέ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λοιπόν πώς ερμηνεύεται αυτή η επιλογή μέσα στο κόρπους της οδηγίας. Επίσης κάτι άλλο το οποίο παρουσιάστηκε εχθές για την εξωτερική πολιτική, για τον εξωτερικό συντονισμό, νομοθεσία για την οποία θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε στοιχεία για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να περιορίσουμε αυτό το χάσμα από το 10% στο 20% της εξοικονόμησης, τι συνέπειες μπορεί να έχει ως προς την εξάρτηση της Ευρώπης από εξωτερικές πηγές ενέργειας και το ισοζύγιο πληρωμών βεβαίως σε οικονομικούς όρους. Πόσα χρήματα θα εξοικονομήσουμε χρήματα δηλαδή τα οποία δεν θα χρειάζεται να δαπανάει η ευρωπαϊκή οικονομία προς τρίτες χώρες για την αγορά ενέργεια, αλλά θα μπορεί να αφιερώσει και να επενδύσει σε ε, θέσει εργασία. Και επίση, μια και βρισκόμαστε σε δυσχερεί οικονομικέ περιόδου, θεωρώ ότι ένα από τα κύρια ζητήματα που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σα είναι το πού ανεβρίσκονται Ε, ελκυστικοί τρόποι προσέλκυσης ε, επενδύσεων. Με την καινοτομία, Φερρυπίν, μπορούμε να πούμε ότι προσελκύουμε μια επένδυση και μετά έχουμε μακροπρόθεσμα ε, πολύ σημαντική εξοικονόμηση κόστους από την ενέργεια, η απόδοση στη δαπάνη. Στην ερώτησή σας όμως, η αγορά ΕΣΚΟ, εξοικονόμησης, δηλαδή αγορά των επιχειρήσεων εξοικονόμησης ενέργειας, έχει πολύ μεγαλύτερη διάδοση και επέκταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια επιχείρηση λέει τι κάνει, κάνει καταβάλει προκαταβολικά το δαπάνη για τον ιδιώτη, για την άλλη επιχείρηση που ενδιαφέρεται να κάνει τη σχετική επένδυση και έχει μερίδιο στη συνέχεια στην απόδοση και τα κέρδη. Έχετε μια τέτοια ιδέα για εξέλιξη αντίστοιχη με αυτή τον ΕΣΚΟ της, ε, των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ θερμά. Να ακούσουμε μόνο δύο-τρει ερωτήσει όμω. Ε, δεν έχουμε περιθώριο για περισσότερε, γιατί τελείω θα είναι και πολύ περίπλοκη η απάντηση που θα δοθεί. Οι ισχυώδει ηγητέ καταρχά, ο καθένα με τη σειρά των ομάδων. Ο κύριο Πίπερ, παρακαλώ. Ναι, καλά κατάλαβα. Είναι η σειρά μου. Και μετά θα έχω και άλλη μια δυνατότητα να μιλήσω. Αν μου δώσετε την υπόσχεση, θα περιοριστώ μόνο σε τρει-τέσσερι ε, ε, ερωτήσεις. Η μέθοδος υπολογισμού που έχετε παρουσιάσει είναι πολύ εντυπωσιακή ως παρουσίαση. Αλλά αν κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά τις επιστημονικές βάσεις πάνω στις οποίες ή τις μεθόδους, τα μοντέλα πάνω στα οποία έχετε στηριχθεί, οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ τουλάχιστον έχω πολλές αμφιβολίες επιλέγεται πάντοτε το σύστημα Primes το οποίο έχει εκτεθεί σε πολύ σημαντικές επίκρισεις προς τη μεθοδολογία του. Πρώτη μου ερώτηση λοιπόν, εσείς ως Επιτροπή δεν έχετε πράγματι κανένα άλλο μοντέλο σε για να ε, διατυπώσετε κατά τρόπο διαφανή αυτούς τους υπολογισμούς και τα μοντέλα. Δεύτερη ερώτηση. Στην ε, πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας που κάνετε την πρόγνωση μέχρι το 2020. Πράγμα το οποίο για μένα είναι εσφαλμένο μεθοδολογικά, αλλά εν αφού κάνετε αυτή την προβολή. Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η καταγραφή εξοικονόμησης, ποιο είναι το έτος αναφοράς με βάση το οποίο λέτε ότι θα έχουμε την εξοικονόμηση στο έτος 2020 με βάση την κατανάλωση του 2007, 8, 10. Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Και επίσης λαμβάνονται υπόψη πρώιμες early actions, πρώιμες δράσεις δηλαδή στους υπολογισμούς σας. Πολλά λοιπόν έχουμε να ε, σημειώσουμε ως παρατηρήσεις σχέση με τη μεθοδολογία που έχει επιλογή. Τρίτος τομέας, για το ενδεχόμενο να μην επιτευχθούν οι στόχοι προτείνεται να επιβάλλεται συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα μέτρα στα ε, κράτη-μέλη που θα πρέπει να ισχύσουν από το 2016 κτλ. Φερρυπίν η Γερμανία. Η Γερμανία έχει ένα εθνικό σχέδιο αποτελεσματικότητας στη χρήση της ενέργειας και φαίνεται ότι θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους που έχουν οριστεί κατά 330, κατά 330% δηλαδή 3,3 φορές. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς μπορεί αυτή η εξοικονόμηση στο 1,5% το οποίο έχετε ορίσει εσείς ως βέλτιστο και ένα ως ε, χείριστο πρέπει να ε, εξισωθεί για τους πάντες. Γιατί δηλαδή θα πρέπει κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα να μειώσει την, ε, την απόδοσή του. Ή γιατί θα πρέπει να έχει την ίδια μεταχείριση με άλλα κράτη τα οποία έχουν λιγότερο καλές επιδόσεις προς την εξοικονόμηση ή λιγότερο καλές μεθόδους επιλέξει. Τελευταίος τομέας, επικουρικότητα, την οποία θα εκθέσω περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι, η πολιτική προσέγγιση λέτε ότι 1,5% ετήσια μπορούμε να επιτύχουμε, μπορεί να μας οδηγήσει σε ε, μείωση ικανοποιητική περισσότερο από ό,τι αν είχαμε την πίεση και την όθηση που μπορεί να προσφέρει η ε, ελεύθερη αγορά. Όμως αυτό σας σε αυτό σας διαψεύδουν κράτη όπως η Γερμανία, η οποία μόνο με τα κριτήρια της αγοράς και τα κίνητρα της αγοράς έχει επιτύχει διπλάσια, τριπλάσια ακόμη ε, βελτίωση σε σχέση με τους στόχους που είχαν προσδιοριστεί. Και εγώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος της ομάδας μου την Κομισιόν για την παρουσία της εδώ στην Επιτροπή μας για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα έχουμε χρόνο βέβαια μπροστά μας για να συζητήσουμε όλα τα σημεία τα οποία τέθησαν. Απλώς ε, σήμερα θα ήθελα να θέσω επιτάπητος ορισμένα προβλήματα σχετικά με αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Όπως γνωρίζετε, η ομάδα μας πάντοτε υποστήριξε να έχουμε ένα δεσμευτικό στόχο. Για να κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό του ποσοστού και στη γραμμή που ανέφερε και ο προλαλής σας, Χρειαζόμαστε μία μεθοδολογία η οποία να είναι αποδεκτή και σωστή για όλα τα, κρά... για όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε μεγάλες αλλαγές. Έχουμε μεγάλες αλλαγές. Το planning... Ay, ya ha Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να διερευνήσουμε άλλους στόχους. Για παράδειγμα, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την ιστορικότητά της τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως αναφέρεται στην οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες. Θα ήθελα να ξέρω πιο συγκεκριμένα τι πιστεύει η Κομισιόν για αυτές τις δύο παραμέτρους και μία δεύτερη ερώτηση θα ακολου... κύριε Πρόεδρε για το θέμα των δημόσιων κτηρίων διότι μας έχουν αναφερθεί προβλήματα σχετικά με τις προθεσμίες οι οποίες είναι πάρα πολύ περιορισμένες δημιουργούν πρόβλημα στα κράτη-μέλη διότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2014 πρέπει να έχουμε μια λίστα των δημοσίων κτηρίων. Κυρίως ε, το πρόβλημα είναι στις χώρες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα αποκεντρωμένη διοίκηση. Η χωροταξική τους ε, διάρθρωση είναι ιδιαίτερα πιο πολύπλοκη και μπορεί να έχουν δυσκολίες. Ε, για να κρατήσουν αυτές τις προθεσμίες. Ρωτώ λοιπόν την Κομισιόν αν υπόψη της τις δυσκολίες των κρατών μελών που έχουν μία πολύπλοκη χωροταξική συγκρότηση. Thank you. Um, I I Στην πρόταση Επιτροπής αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς το πόσο επίγον και σοβαρό είναι το πρόβλημα που έχουμε η κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης. Και είναι απολύτως απαραίτητο και για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να κάνουν εξοικονομήσεις ε, πόρων ως προς τους ε, πόρους που χρησιμοποιούν. Χρειάζεται δηλαδή αυτή η εξοικονόμηση. Κατά αυτό τους 368 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμο πετρελαίου τουλάχιστον. Αυτό που βλέπω λοιπόν είναι ότι μάλλον δεν είναι αυτό το σχέδιο τόσο φιλόδοξο όσο θα έπρεπε να είναι ή όσο φαινόταν ότι θα είναι αρχικά και ίσως να μην προσφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα λόγω λήψης φιλοδοξία. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή εάν μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να παραδεχθεί ότι αυτή η επιλογή δεν είναι επαρκής και ότι κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να αλλάξουν και συμπεριφορά αντιλαμβανόμενα την σημασία της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Το δεύτερο θέμα είναι το χρονοδιάγραμμα και πάλι έχουμε να κάνουμε με την, έχει να κάνει εδώ με τη σημασία του να αντιληφθούμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να συμβεί και ότι δεν αποτελεί μόνο μια φιλοδοξία επιχάρτου. Και εδώ θέση έχει η Επιτροπή με τις προβλέψεις της για το τι θα επιτύχουν τα, τα κράτη του 2014, νύβια τα σχήρα της δηλαδή, γιατί παραπέμπει το θέμα στην προσεχή Επιτροπή και εκεί οι προτάσεις θα κατατεθούν κάπου το 2015-2016, άρα σίγουρα θα έχουμε το χρόνο για να φτάσουμε στο 2020 με επαρκή αποτελέσματα. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να συμβεί ουσιαστικά και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το επιτύχουμε. Και θα ήθελα η Επιτροπή να μιλήσει πιο καθαρά και σε λεπτομέρειες ως προς το συσχετισμό με το σύστημα των ανταλλαγών εκπομπών, το ETS λέτε ότι θα καταβάλει κάθε προσοχή, θα παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή κτλ. Μα εδώ έχουμε ένα κάνουμε ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει το κάθε τμήμα, η κάθε διεύθυνση να δουλέψει σε στενή συνεργασία με όλες τις άλλες. Πρόκειται για κάτι το θετικό. Και πρέπει να φροντίσουμε να μειώσουμε το όριο ως προς εκπομπές για να έχουμε την ε, βέλτιστη δυνατή απόδοση. Άρα ίσως να μην έχουμε αρκετά ε, αποτελέσματα ε, στην ε, ώρα που χρειάζεται να τα έχουμε. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ρόιλ. Παρακαλώ, κυρία Φόρτ. Παρακαλώ. Μερικά σύντομα σχόλια μόνο. Ασφαλώς και οι λοιποί συνάδελφοι σκιώδης συντηνιστές θα έχουν ε, λάβει στο ηλεκτρονικό του μέτρη μέτρητα μηνύματα από διάφορους είτε πρόκειται για τοπικέ αρχές, μικρέ μεσέ επιχειρήσει, μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιώτες που θεωρούν ότι έχουν κάποιες προτάσεις και μπορούν να βοηθήσουν στην διατύπωση των όρων και των ε, μέτρων ε, Τώρα που έχουμε το κείμενο σας μπορούμε να συγκρίνουμε στη σχέση με αυτά που έχουν ήδη προταθεί. Ασφαλώς η Φιώνα αυτό που θέλει να πει είναι ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργεια για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Εσείς όμως είχατε προσδιορίσει για το 2010 την ε, περικοπή ενεργειών, ενέργειας και όχι εξοικονόμησης. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μιλάμε για εξοικονόμηση και όχι για περικοπές. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι, όπως σημανθήκε νωρίτερα, να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία για λόγους εταιρικούς έχουν κάνει ε, μια δική τους προσπάθεια. Φερρυπίν, ε, στην ε, Βρετανία είχαμε ένα θέμα το οποίο προχώρησε πολύ σε ευρύ βαθμό ε, με την μόνωση, θερμομόνωση των κατοικιών, ε, στην Ιταλία με τα συστήματα φωτισμού. Έχουν αναλυφθεί δηλαδή μέτρα σε ορισμένα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσετε να μην είναι τα μέτρα που θα επιβάλλετε ή που θα ε, διατυπώσετε εσείς υπερβολικά δεσμευτικά. έτσι ώστε να μην επιβληθούν ε, μέτρα ή λύσεις που θα οδηγήσουν σε αντιπαραγωγικές ε, αντιδράσεις τους ε, ανθρώπους. Δηλαδή να πάει κανείς να κατασκευάσει μια μονάδα κάπου μόνο και μόνο γιατί περιμένει ότι θα αποκομίσει όφελος από κάποια από τα μέτρα ενώ στην ουσία δεν έχει αυτό οικονομικό και ε, περιβαλλοντικό ε, αντίκτυπο. Θετικό αντίκτυπο δηλαδή. Αυτά πρέπει να δούμε και βέβαια θα τα εξετάσουμε τι προτάσεις και θα καταθέσουμε το τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Ρόιλ. τώρα παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους βουλευτές. Κύριε Τσουρμές, ναι, έχετε δίκιο ότι το άρθρο 6 μιλάει για το ίμιση των ε, επιδιωκόμενων στόχων Η ανάλυση, ωστόσο, είναι συνεπής και παραμένει μέσα στο 6-9 το τωρινό όπου αφού περιγράφηκαν ε, οι υποχρεώσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, σημειώνεται ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, προχωρήσουν σε, επιπλέον, σε τύπος επιπλέον στόχους ε, που θα είναι ισοδύναμοι ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας με αυτούς της παραγράφου 1 σχέση με τους δυτικούς πελάτες. Άρα δεν έχουμε αντίφαση εδώ. Θα υπάρξει φυσικά σημαντικός αντίκτυπος ως προς την εξάρτηση σε ενέργεια. Δηλαδή το ένα δεύτερο τουλάχιστον της εξοικονόμηση θα είναι εξοικονόμηση από εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Οι πληρωμές σε οικονομικούς όρους θα σημάνουν εξοικονόμηση 18 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 2020 περίπου, ίσως με κάπως συντηρητική αξιολόγηση. Συμφωνούμε με τον κύριο Τουρμές ε, για την ανάγκη να προσελκυθεί και ιδιωτικό κεφάλαιο. Η αγορά η σχετική των ΗΠΑ είναι 10 με 20 φορές μεγαλύτερη από αυτές της ε, Ευρώπης και μάλιστα της Γερμανίας, γιατί η να κράτη είναι ακόμη πιο πίσω. Και μάλιστα αυτές οι επιχειρήσεις για τις οποίες μιλήσατε είναι μια καταπληκτική ιδέα, διότι προκαταβάλουν το κόστος της εξοικονόμησης ενέργειας, της πιο αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας, που έχει φυσικά πολύ μεγάλη απόδοση, αλλά που δεν διαθέτει ο κάθε ιδιώτης, το κάθε νοικοκυριό, και μετά από την εξοικονόμηση ενέργειας αποκομίζουν αυτές οι ε, εταιρείε την απόδοση και το κέρδος τους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε και για την Ευρώπη. Αυτές οι ΕΣΚΟ είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα λύση και από το δημόσιο τομέα πρέπει να τις ε, προωθήσουμε πιστεύω, αν και κυρίως ε, αναπτύσσουν δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει λοιπόν η εξαγορά και η ανακαίνιση κτηρίων στον δημόσιο τομέα να αποτελέσει μια ευκαιρία για ανάπτυξη επιχειρήσεων τύπου ΕΣΚΟ και στην Ευρώπη. Για τον κύριο Πίπερ συμφωνώ ότι πολλή δουλειά πρέπει να γίνει ακόμη για να βελτιωθούν τα διάφορα μοντέλα και η αξιολόγηση αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας. Εμείς ακολουθούμε μοντέλα τα οποία προκύπτουν από την παράδοση της προσφοράς, της προμήθειας σε ενέργεια και ζητούμε από τον καταναλωτή να δώσει στοιχεία ε, που του είναι λιγότερο αυτονόητα από αυτά της προμήθειας. Εάν όμως ορίσουμε δεσμευτικούς στόχους, πάλι θα πρέπει εγώ να ζητήσω υπερασπιζόμενος μέχρι τελευταία δρανίδα του αίματός μου τα μέτρα αυτά τα οποία έχουμε προτείνει. Γιατί αν ξεφύγουν από τα μοντέλα τα μέτρα, τα πρότυπα είτε είναι της Γερμανίας, είτε είναι της Ρουμανίας, της Ιταλίας, φύχη ψή, ωμέγα, δεν έχουν ε, για μας τα μέτρα τα οποία προτείνουμε εμείς διαφέρουν από τα μέτρα των κρατών μελών, διότι δεν έχουν δεσμευτικούς στόχους. Και αν επανέλθουμε με πρόταση για δεσμευτικούς στόχους του 2014, θα είναι απαραίτητο προηγουμένω να έχουμε βελτιώσει τα μοντέλα μας. Για την πρόταση αυτή, λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι ότι εισαγάγαμε ήδη τι αλλαγέ στην προσέγγιση primes που καθιστούν την ε, το μοντέλο προς τη συμπεριφορά του καταναλωτή κάπως πιο λεπτό, βλέπει πιο πολλές λεπτομέρειες και έχουμε κάνει και αντιπαραβολή με το E3ME. Ε, e. Και χωρίς να είμαστε 100% πεισμένοι ότι έχουμε το βέλτιστο δυνατό μοντέλο, βλέπουμε ότι έχουμε πιάσει μια γκάμα αρκετά καλή αποτελεσμάτων, αρκετά αξιόπιστη πρώιμη δράση, αν θα αντιλάβουμε υπόψη. Βεβαίω, αυτό που ζητούμε από τα κράτη-μέλη είναι να προσδιορίσουν τα ίδια ένα στόχο για το 2020. λαμβανομένων υπόψη και των νέων μέτρων που θα εισαχθούν. Και έτσι τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν αναλάβει πρώιμη δράση, δράση, θα είναι εκείνα τα οποία θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή την εξέλιξη. Και φαντάζομαι ότι και εκείνα που έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό θα ωφεληθούν περισσότερο. Και ασφαλώς θα φτάσει στο 20% ελπίζουμε όλα μαζί τα κράτη. Ιδάλω το 2014 θα επανέλθουμε με μια πρόταση για δεσμευτικά μέτρα. Για το 1,5% του άρθρου 6 που οδηγεί, όπως είπε ο κύριος Τουρμές, το άρθρο 6 σε σοβαρές ε, εξοικονομήσεις. Είναι πολύ φιλόδοξο το ποσοστό αυτό. Τα στοιχεία όμως που έχουμε δείχνουν ότι αυτό είναι ο στόχος και το επιτυγχανόμενο αποτέλεσμα σε ανεπτυγμένες οικονομίες αλλού. Άρα, αν αυτό εννοείται με την ερώτησή σας, χώρες με υψηλότερο δυναμικό από άλλες, αλλά και χώρες με όχι τόσο μεγάλο δυναμικό, έχουν δυσκολία θα έχουν ε, ενδεχομένω όχι τόσο μεγάλη ευκολία προ την επίτευξη αυτών των χρόνων αυτών. Για την κυρία Μαντουρέλ. Εν μέρη επανέρχομαι με την απάντηση προς τον κύριο Πίπερ ότι δηλαδή τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε εσείς έχουν μεγάλη σημασία εάν εξετάσουμε τις πιθανές εξελίξεις ενός συνόλου εθνικών στόχων σε εθνικό επίπεδο. Θα ήταν σημαντικό φυσικά να αναλυφθεί ε, πρόορη δράση, αλλά και να προσδιοριστούν τάσεις ε, και ένταση ενέργεια. Ως προς τα μέτρα περί καταγραφής και απόδοσης ε, λογαριασμών ή εκθέσεων, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να καταγράψουν όχι μόνο τάσεις σε χρήση ενέργειας, αλλά και τάσεις σε ένταση ενέργειας ανατομέα, έτσι ώστε η αξιολόγησή μας να μην λέει μόνο η Ισπανία έχει φέρει πίν ε, μεγαλύτερη χρήση ενέργειας στις μεταφορές, αλλά να έχουμε και την εξήγηση ότι οι μεταφορέ χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια γιατί έχει αναπτυχθεί η οικονομία και άρα υπάρχουν περισσότερε μεταφορέ ή γιατί δεν είναι τόσο καλή η αξιοποίηση ενέργεια. Αυτό είναι ε, πολύ σημαντικό, όπω λέτε κι εσεί, να καταγράφετε. Ω προ το χρονοδιάγραμμα για τι απογραφέ αυτέ, η οδηγία για την αξιολόγηση ε, ενεργειακής απόδοσης κτηρίων απαιτεί δημόσια κτίρια να ε, λαμβάνουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Βέβαια, οι μικρότερες ομάδες κτηρίων που καλύπτονται από την παρούσα πρόταση που μιλούν για 2015 ή μέχρι το 2014 δεν αποτελούν ε, μία σοβαρή καινοτομία, δεν ε, ε, ορίζουμε τίποτα το καινούριο, απλώς στηριζόμαστε και αναπτύσσουμε την υφιστάμενη πρόταση. Για την κυρία Χολ, ασφαλώς συμφωνώ ότι χρειάζεται αυτή η προσπάθεια να δώσει καρπούς σε δεδομένη οικονομική κρίση. Και ακριβώς σε περίοδο οικονομικής κρίσης δεν έχει νόημα να εκλείεται η θερμότητα από τα σπίτια που προσπαθούμε να θερμάνουμε και να διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Σημασία έχει με τέτοια περίοδο να εξοικονομούμε αυτή την ενέργεια, να έχουμε κλειστά παράθυρα και να την αξιοποιούμε τη θερμότητα κάπως ε, αλλιώς ε, να εξοικονομούμε χρήματα και να στηρίζουμε τη βιομηχανία ε, για παραγωγή προϊόντων πιο αξιόπιστων, πιο αποτελεσματικών καλύτερα προς την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, θεραπείν, λέβητες, με καλύτερη αποτελεσματικότητα ή παράθυρα ε, με καλύτερη θερμομόνωση. Όλα αυτά, όπως προτείνει και ο κύριος Τουρμές, μπορούν να προχωρήσουν μέσα από ε, συνεργασία και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και, μέσα από το, και να στηριχθούν από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όσον αφορά την διασύνδεση με το ETS, αφού έχουμε δύο διαφορετικά μοντέλα που από τα οποία προκύπτουν διαφορετικές απαντήσεις, από τον οποίων το ένα λέει δεν υπάρχει πρόβλημα και το άλλο επισημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, θεωρήσαμε ότι στην παρούσα πρόταση δεν ήταν σκόπιμο να μιλήσουμε για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά θεωρούσαμε ότι είναι σκοπιμότερο να συνεχίσουμε την αξιολόγηση του κατά πόσον θα προκύψει το πρόβλημα αυτό. Για δε την κυρία Φόρντ, Προσπαθήσαμε να αναγνωρίσουμε και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και να ε, διαπιστώσουμε ότι όντως έχουμε να κάνουμε εγγενείς διαφορές, με τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ε, χρησιμοποιεί την ενέργεια ή ενημερώνεται, ζητεί και λαμβάνει την πληροφόρηση. Ε, άρα λοιπόν θα αφήσουμε επαρκές πεδίο ε, δράσεις στα κράτη-μέλη. Δεν θα προχωρήσουμε σε πλήρη εναρμόνιση. Ο κύριος Ρόιλ, ευχαριστώ πολύ. Αν τυχόν δεν έχουν δοθεί ε, απαντήσει επαρκή, ε, επαναλάβετε τις ερωτήσεις σα, αλλά πρέπει να προχωρήσω τώρα. Ένσω. εσείς παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τόσο από οι συνάδελφοι. Μία πτυχή μόνο, που είναι πολύ σημαντική. και είναι η αποτελεσματικότητα σε ενέργεια των κτηρίων. 44% της χρήσης των ε, κτηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αφιερωμένο στα, ε, προέρχεται μάλλον από τα κτίρια και το 19% των εκπομπών αερίων ε, θερμοκηπίου επίσης προέρχεται από κτίρια. Μία πτυχή λοιπόν που θα ήθελα να αναφέρω στην οδηγία κάνουμε, γίνεται επιστολή αναφορά στα δημόσια κτίρια. Ναι. Λέγεται όμως ταυτόχρονα ότι τα δημόσια κτίρια αποτελούν ε, ε παρουσιάζουν κατά 3% ανάγκη για ανακαίνιση. Αλλά στο συνολικό ε, αριθμό δημοσιο... Ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δημόσια είναι πολύ λίγα. Τα περισσότερα κτίρια είναι σε χέρια ιδιωτών, ιδιωτικά. Άρα για να δράσουμε, για να βρούμε έναν τρόπο να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα στην ενεργειακή χρήση αυτών των κτίριων, θα πρέπει να κοιτάξουμε τα ιδιωτικά κτίρια. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε κράτος μέλος έχει χαρακτηριστικά δικά του, όπως άλλωστε δείχνει και η πρόταση της Επιτροπής. Στη Ρουμανία Φερρυπίν 19% των κτίριων είναι κτίρια που βρίσκονται σε ιδιοκαθήκηση, δηλαδή ανήκουν στον ένικο. Η Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει το κόστος τέτοιων κτιρίων να κατανεμηθεί μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενίκου. Εδώ όμως, στη δική μας περίπτωση, δεν θα έχει εφαρμογή, γιατί 19% των κτιρίων ε, χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση. Πώς μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση της Ρουμανίας να υποχρεώσει έναν ιδιοκτήτη κτηρίου που διαμένει σε αυτό να αναλάβει ολόκληρο το κόστος της ανακαίνησης του κτηρίου δεδομένου ότι το μέσο εισόδημα στη Ρουμανία είναι κάτω από 400 ευρώ και η μέση σύνταξη κάτω από 180 ευρώ. Άρα θα πρέπει να βρούμε ε, κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Επιδοσφαλός ε, για να στηρίξουμε με δάνεια ή επιδοτήσεις τους ίδιοκτες αυτούς που θα θέλουν να ε, τα κτίρια τους και να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφος Γκέρεκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπερδεύουμε την αποτελεσματικότητα με την, εξοικονόμηση. Η εξοικονόμηση αποτελεί μια λειτουργία της αποτελεσματικότητας. Η Κομισιόν μπερδεύει τα πράγματα, τα προστεύει ιδιαίτερα μάλλον καλύτερα, διότι και τα δύο τα βάζει στο ίδιο επίπεδο. Οπότε τι θα συμβεί. Οι κυβερνήσεις θα περιοριστούν απλώς να κλείνουν τον διακόπτη αντί να αναζητούν την πραγματική αποτελεσματικότητα που σημαίνει μόνωση, μείωση της σπατάλης των διαφυγών ενέργειας, αλλαγή των συστημάτων. Πώς την εννοεί όμως την αποτελεσματικότητα η Κομίσιον διότι αν για την Κομισιόν η αποτελεσματικότητα είναι ένα ακαθάριστο, ένα μεικτό μάλλον, μια, μια μεικτή εξοικονόμηση για την κάθε χώρα, δηλαδή συνδυασμός εξοικονόμησης και αποτελεσματικότητας με δίκτυ κατά κεφαλήνα. Στην Πολωνία όμως τι σημαίνει το την η κατακεφαλίνα κατανάλωση. Ας πούμε στην Πολωνία καταναλώνουμε 10 φορές λιγότερο από ό,τι στη Γερμανία. Και αν πάρουμε την μεικτή ε, τιμή τότε εμείς μειώνουμε την, την ενεργειακή ε, την ενεργειακή κατακεφαλήν εξοικονόμηση τότε φύγουμε τις πιο φτωχές χώρες τύπου δηλαδή Ρωμανία και, Ρωμανία και Πολωνία. Δηλαδή αποτελεσματικότητα πάνω από το, 20% κατακεφαλήν αλλά αυξάνοντας για τις στοχότερες χώρες, π.χ. για την Πολωνία, ένα συγκεκριμένο ποσοστό για την, για την κατανάλωση, τότε αλλάζει το πράγμα αλλά αλλιώς ε, πλήττουμε τις πιο φτωχές χώρες. Πρωτογενής ενέργεια. Πολύ ωραίος όρος. Φύγουμε τις, ε, όλες τις ε, πηγές ενέργειας. Και μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τεχνικές πρόοδους και προσαρμογές. Ας μου το εξηγήσει η Κομισιόν τι εννοεί ως πρωτογενή εξοικονόμηση. Εμείς είχαμε ορίσει στο παρελθόν ένα κλιματικό πακέτο και τότε άμα όταν το ορίζαμε είχαμε μιλήσει και για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα σήμερα θα είχαμε και τις πρώτες οικονομίες. Τώρα, επειδή το πακέτο θεωρεί ότι τα ορυκτά τα κάψιμα θα χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον. Και θέλω να ρωτήσω, άμα θέλουμε εμείς αποτελεσματικότητα 120%, εγώ δεν μπορώ να ανοίξω κανένα νέο εργοστάσιο ε, παραγωγής ενέργειας χωρίς ε, να έχω τις, ε, τα ETS μπροστά μου. Ο κύριος Βανίστερο, εγώ θα είχα δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η εξής. Εμείς στην τοποθέτησή μας, στη θέση μας μάλλον είχαμε πει πρώτα ότι τα κράτη-μέλη έπρεπε να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα και μετά θα γινόταν συζήτηση στο πλαίσιο της Κομισιόν. Αλλά δεν ακούω πια τίποτα. Τι κάνει η Κομισιόν για την πρώτη φάση και για την ρύθμιση. Σίγουρα Έχουμε ενεργεια... Έχουμε τεχνικά επιχειρήματα, τα οποία όμως δεν με πείθουν και πολύ. Και υπάρχει και κάτι άλλο που δεν με πείθει. Λέμε, ας πούμε, στη Ρουμανία χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρηματοδότηση. Αλλά, αγαπητοί φίλοι, έχουμε τα διαρθρωτικά ταμεία και μάλιστα προσαρμόσαμε και τον κανονισμό που λέει ότι το 7% των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Η Ρουμανία δεν χρησιμοποίησε φράγκο από, αυτά τα κονδύλια. Η Γαλλία ναι. Εγώ διάβασα το δημοσιονομικό πλαίσιο και λέει ότι το ποσοστό που θα χρειαστεί για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα θα πρέπει να ανέλθει στο 10%. Αλλά δεν έγινε πραγματική συζήτηση ούτε καν στο πλαίσιο της Επιτροπής. Για την ε, διαχείριση πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση και να δούμε και ποιο ε, μοντέλο θα ακολουθήσουμε το πιο αποτελεσματικό. Εμείς μιλάμε ένα σωρό για ρύθμιση, απορρίθμιση κτλ. Αλλά αυτό δεν με πείθει. Ο κύριος Βέμπερ. Και εγώ δεν θέλω να επαναλάβω όλες τις εύστοχες ερωτήσεις των συναδέλφων. Εγώ θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία της παρουσίας της Επιτροπής για να ρωτήσω κάτι το συγκεκριμένο και που αφορά στη ανάπτυξη των ευφυών δικτύων, τα smart grids που επιτρέπουν μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα στην Ένωση. Όμως η εξέλιξη των smart grid βρίσκεται σε εμβριακό στάδιο στην Ευρώπη το θέμα της διαλειτουργικότητας αλλά ε, και το δελτίο όρων εφαρμογής δεν υφίσταται ακόμα. Πρέπει λοιπόν εμείς να ορίσουμε τους κανόνες. Ορίζονται βέβαια, θα οριστούν μέχρι τα τέλη του 2012. Εγώ είμαι μέλος της, Κίνας, ε, της Αντιπροσωπείας Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και 270 εκατομμύρια ευρώ, 2 δις η Ιωάννα μέχρι το 2005 θα αξιοποιήσει, ε, θα τα επενδύσει για τα smart grids και μέχρι το 2020 η Κίνα θα είναι έτοιμη. Εγγένιασαν και πρότεινο στη Σανγκάη ένα κέντρο έρευνας για τα smart grids. Αυτό τι σημαίνει, όπως πολλοί θα φοβούμε, ότι, τους, ότι ο ορισμός των κανόνων για την βιομηχανία ηλεκτρικής, ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι, οι κανόνες λοιπόν ορίζονται στην Κίνα τι κάνει λοιπόν η Κομισιόν ούτως ώστε να επιβάλλει τους ευρωπαϊκούς κανόνες στη διεθνή αγορά ούτως ώστε να μην καπελωθούμε αύριο από τους ανταγωνιστές μας ο κύριος Μπρεζίνα Συμμερίζομαι τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Θα ήθελα όμως να επανέλθω σε ένα γενικό θέμα. Ρώτησα την Επιτροπή εάν έχει συμπεριλάβει στους συλλογισμούς της ε, ένα παράδοξο οικονομικό φαινόμενο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο συνάδελφος Κίρεκ και ότι ε, συγχαίουμε εδώ δύο πράγματα, την απόδοση της ενέργειας με τις ε, γενικές εξοικονομήσεις ε, και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Όσον αφορά την μελέτη επιπτώσεων για την, ε, που αφορά την έκθεση αυτή, ε, δεν με έχει πείσει ένα πράγμα. ότι δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη εξοικονομήσεις στον τομέα των μεταφορών. Και γενικά θα ήθελα να πω ότι ε, εδώ υπάρχουν ε, υπερβολικά πολλά αναγκαστικά μέτρα. Εάν όμως ε, θέλουμε να έχουμε κεφάλαιο, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα μέτρα που σχετίζονται με τις τιμές. Όταν κοιτώ αυτό το σχέδιο, ντρέπομαι όταν σκέφτομαι τις τσεχικές επιχειρήσεις και ότι ε, κάθε επιχείρηση θα πρέπει ε, να κάνει έναν ε, απολογισμό ενέργειας. Κάτι τέτοιο υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Κάθε επιχείρηση θέλει να εξοικονομήσει χρήματα σε όλους τους τομείς και γι' αυτό πιστεύω ότι τέτοια νομοθεσία δεν είναι καλή για την μελλοντική εξοικονόμηση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, θα ήθελα τότε να δώσω τον ε, λόγο στον ομιλητή για να απαντήσει. Και μετά θα έχουμε τον επόμενο κύριο ερωτήσεων. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Ε, ως απάντηση στον κύριο Ένσο, να πω ότι έχετε δίκαιο που επικεντρώνεστε στο θέμα αυτό ε, των κτηρίων και είναι κάτι που ξεπερνάει ε, το 2020. Θα πρέπει να κοιτάξουμε το 2050 και αν θέλουμε να πλησιάσουμε στο και τους στόχους μας θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Την ε, ενεργειακή ε, ε, ανακαίνιση των κτηρίων δημοσίων και ιδιωτικών και Έχετε δίκιο ότι το να λέμε στον κόσμο ότι θα πρέπει να ε, ανακαινήσει τα κτίρια, να επισκευάσει τα κτίρια, ε, αυτό σίγουρα δεν επίπτει στην ε, δημοκρατική διαδικασία την οποία ακολουθούμε. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ήδη έχουμε κάποιες απαιτήσει ε, στην σχετική οδηγία που λέει ότι κατά την ανακαίνιση των κτηρίων αυτή θα πρέπει να γίνεται ώστε τα κτίρια να γίνονται ενεργειακά αποδοτικά. Έχουμε λοιπόν έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ότι όταν γίνεται η ανακαίνιση, τα κτίρια που θα προκύπτουν είναι αυτά που θέλουμε. Το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να ε, επιταχύνουμε την ε, ανακαίνιση. Ε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο δημόσιο τομέα και για να δείξουμε ότι είναι δυνατή η επιτάχυνση, για να δείξουμε ότι τα οικονομικά ωφέλη είναι σημαντικά και για να δημιουργήσουμε μια αγορά ε, και για τους ε, εξειδικευμένους εργάτες που ε, ελπίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα εξαπλωθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν αρκεί όμως για να πετύχουμε την επιτάχυνση που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2050, είναι όμως ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον, η εμπειρία χωρών όπως είναι ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία μας δείχνουν ότι όταν υπάρχει υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας ε, από την πλευρά της, του τομέα ε, που προμηθεύει την ενέργεια, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με βελτίωση των κτηρίων. Αυτός είναι ένας ελκυστικός τρόπος να γίνει αυτό, δεν είναι πάντα βέβαια ο προτιμητέος. Ε, και τέλος, ο κύριος ε, Φανίστερόι αναφέρθηκε και στο πολιετές ε, ενεργειακό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί μέρος της προσέγγισης της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου. Ε, που παρουσιάστηκε στην ανακοίνωση της 24 Ιουνίου, ε, που λέει ότι ε, μεγάλο μέρος των ταμείων σύγκληση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Αυτό βέβαια θα συζητηθεί στη βάση ξεχωριστή νομοθετική πρόταση. Σε απάντηση στον κύριο Γκίρεκ, να πω ότι και πάλι δεν ε, προτείνουμε εδώ ε, δεσμευτικό στόχο για την Πολωνία ή για άλλο κράτος μέλος. Αυτό που προτείνουμε εδώ είναι μία σειρά δεσμευτικών μέτρων τα οποία θα ε, οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το στόχο που έχει θέσει, ο οποίος είναι 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με ε, την ε, παρούσα κατανάλωση. Αλλά αυτόν τον στόχο δεν τον μετατρέπουμε σε εθνικούς στόχους. Ζητάμε από το κάθε κράτος μέλος, από τη στιγμή που θα έχει υιοθετηθεί η οδηγία, να εντοπίσει, να θέσει τους δικούς του εθνικούς στόχους. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι οι πολωνικές αρχές θα λάβουν ε, υπόψη αυτά που μας αναφέρατε κατά τον καθορισμό των στόχων της. Αλλά στο κείμενο που παρουσιάσαμε εμείς ε, δεν ε, ε, περιορίζουμε τις επιλογές της Πολωνίας. Θα πρέπει η Πολωνία να θέσει τους στόχους λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα δεσμευτικά μέτρα θα μειώσουν την κατανάλωση με αυτήν που θα ήταν χωρίς τη λήψη μέτρων. Συμφωνούμε ότι είναι καλό να εργαζόμαστε πάνω στον πρωτογενή ενεργειακό τομέα, επιτρέποντας έτσι να ε, εξοικονομήσουμε χρήματα αυξάνοντας την απόδοση για την ε, παραγωγή ενέργειας και θέρμανσης ε, καθώς και κατά την κατανάλωση. Το CCS ήταν η τρίτη σας ερώτηση. Ε, το αναγνωρίζουμε αυτό και θα θέλαμε πολύ να δούμε ε, ανάπτυξη του CCS. Ε, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά αυτό το λαμβάνουμε υπόψη στις προτάσεις μας εδώ πέρα. Ε, δεν θεωρούμε λοιπόν ε, ότι ε, αυτό θα είναι εμπόδιο. Κύριε Φανίστελ Ρόι, τι θα κάνει η Κομισιόν κατά την πρώτη αυτή φάση που θα οδηγήσει στην πιθανή πρόταση δεσμευτικών, μέτρων, δεσμευτικών στόχων. Όπως σας είπα, το πρώτο είναι ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να θέσει εθνικούς στόχους. Αυτό θα ζητηθεί από τα κράτη-μέλη στις αρχές του 2013. Και όπως είπατε κύριε Νίστελ Ρόι, Καταρχήν ε, θα ε, κοιτάξουμε όλους τους εθνικούς στόχους και να δούμε εάν ε, το άθροισμά τους θα είναι η εξοικονόμηση κατά 20%. Δεύτερον θα εξετάσουμε τα εθνικά σχέδια για να δούμε εάν εάν είναι εφικτά. Δηλαδή, αν τα κράτη-μέλη θέλουν να πετύχουν μείωση κατά 20%, τα μέτρα αυτά αρκούν για να το πετύχουν αυτό. θα κοιτάξουμε με θετικό μάτι τις προτάσεις. Και τρίτον, ε, τι ε, θα γίνει παράλληλα από τώρα μέχρι την αξιολόγηση αυτή που σας ανέφερα, ε, τις αρχές του 2014 δηλαδή. Για, για παράδειγμα, την εισαγωγή μέτρων οικολογικού σχεδιασμού, για παράδειγμα. Και τέταρτον, θα εξετάσουμε ε, ποια θα είναι τα αποτελέσματα της οδηγίας αυτής ε, στην ε, τελική της μορφή. Θα είναι λοιπόν πολύ η ευρεία θα είναι πολύ ευρεία η αξιολόγηση που θα κάνουμε και θα γίνει με βάση τα μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Βέμπερ ερώτησε σχετικά με τα FE δίκτυα, τα smart grids. Η πρόταση αυτή κατά κάποιον τρόπο καλύπτει τα smart grids. Εμείς υποθέτουμε ότι θα έχουμε ένα FES σύστημα και λέμε στον κόσμο ότι οι μετρητές που θα έχουν στα σπίτια τους θα τους επιτρέπουν να ε, ε, ωφεληθούν από τα ε, FE δίκτυα, τα smart grids. Όλα αυτά προϋποθέτουν τα έξυπνα δίκτυα και θα υποβάλουμε πρόσθετες προτάσεις στα πλαίσια του πακέτου υποδομής. Ε, θα προτιμούσα να μην ε, απαντήσω στην ερώτησή σας τώρα, να περιμένετε τη συζήτηση που θα γίνει στο πλαίσιο αυτό, διότι θεωρούμε ότι είναι παράλληλες οι προτάσεις αυτές και ε, εξαρτώνται από και εξαρτώμαστε, εξαρτάται η επιτυχία της συγκεκριμένης πρότασης από την άλλη. Τέλος, στον κύριο Πρεζίνα να απαντήσω. ότι έχετε δίκιο ότι δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες στην μελέτη επιπτώσεων ούτε στην πρόταση με τον ε, τομέα μεταφορών όπου υπάρχει ε, μεγάλη δυνατότητα εξοικονόμησης διότι η Λευκή Βίβλωση για τις μεταφορές που αφορά τις μεταφορές μέχρι το 2015 είναι παράλληλο έργο που προβλέπει εξοικονόμηση νομίζω 65 τόνων πετρελαίου από τον ε, ε, τομέα μεταφορών. Για να πετύχουμε το στόχο του 20% ε, χρειαζόμαστε και την εξοικονόμηση αυτή. Ε, είμαι βέβαιος λοιπόν ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για να επιτευχθεί και αυτός ο στόχος. Και συμφωνούμε μαζί σας ότι αν κοιτάξουμε το συνολικό παρόναμα της ενέργειας, ο βιομηχανικός τομέας έχει ε, κάνει, ε, έχει πετύχει τα περισσότερα μέχρι τώρα και ε, εκεί απομένουν λιγότερα να γίνουν. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης στα κτίρια, στην προμήθεια ενέργειας, στις μεταφορές από ότι στον βιομηχανικό τομέα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε να υπάρχει κάποια δυνατότητα εξοικονόμησης στον βιομηχανικό τομέα. Οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν ε, ένα σχέδιο ενεργειακής απόδοσης ε, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, ενώ ε, τα άλλα, οι άλλες επιχειρήσεις θα πρέπει να το κάνουν. Και για το παράδοξο που μιλήσατε, λυπάμαι, δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφος Τόμσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Η ε, οδηγία για την ενεργειακή απόδοση είναι πολύ σημαντικό θέμα ε, για το οποίο ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας την άνοιξη του 2012. Οι ε, παρούσες εκτιμήσεις ε, δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται καθόλου να πετύχει τους ε, στόχους της για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέχρι το 2020. Με τις παρούσες εκτιμήσεις θα πετύχουμε μόνο το 1 τρίτο αυτού και αυτό βέβαια είναι απαράδεκτο τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι η απόδοση τη ενέργεια είναι ο φθηνότερο τρόπο να εξοικονομήσουμε χρήματα. Είναι σαν να λέμε τα φρούτα που κρέμονται χαμηλά στο δέντρο, που είναι πιο εύκολο να τα κόψουμε. Η ενεργειακή απόδοση είναι ένα πράγμα, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας, όπως είπε ο κύριος Συγκύριακ, είναι διαφορετικό. Ε, εάν όμως θέλουμε να πετύχουμε μείωση της ε, κατανάλωσης, ε, σημαντικό είναι να καταβάλουμε προσπάθειες και στους δύο αυτούς τομείς. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν έχει ε, πολύ καλά στοιχεία σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Ε, επικεντρώνεται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, το οποίο είναι θετικό. Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, δεν καταλαβαίνω το θέμα των δεσμευτικών στόχων. 9 Μαρτίου του 2007... Παρασκευή πρωί υπόθηκε ότι έχουμε, η, η κυρία Μέρκελ είπε ότι ε, στο Συμβούλιο αποφασίσαμε σχετικά με δεσμευτικού στόχους ε, για την ε, οδηγία για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας. Και ποιο ήταν το μήνυμά τη, Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα προς τη βιομηχανία, διότι η βιομηχανία δεν θα επενδύσει εάν δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι. Και γνωρίζουμε από όλε ε, τις εμπειρίες μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όταν δεν υπάρχουν ε, δεσμευτικοί στόχοι και το βλέπουμε αυτό και τώρα που μιλάμε για την απόδοση της ενέργειας και σε προηγούμενες οδηγίες είδαμε ότι δεν βλέπουμε πλήρως των στόχων όταν δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι. Και γι' αυτό θα πρέπει να στείλουμε στην βιομηχανία το μήνυμα χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους και γι' αυτό θα πρέπει η εξοικονόμηση ενέργειας να είναι υποχρεωτική. Ξέρω ότι η συντηρητική φιλελεύθερη κυβέρνηση της Δανίας το καλοκαίρι του 2008 ε, κατάφερε να ε, βρει τη στήριξη του συνολικού κοινοβουλίου από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά ε, στέλνοντας επιστολή στην Κομισιόν που έλεγε ότι έχουμε πολύ καλές εμπειρίες στην στη Δανία, όπου έχει αυξηθεί το ΑΕΠ μας κατά 30% τα τελευταία 20 ε, χρόνια, ενώ η κατανάλωση ενέργειας κατά 12% επειδή έχουμε, δημιουργήσαμε πριν 30 χρόνια ένα πολύ σωστό πρότυπο. Ε, αλλά ε, η απάντηση ήταν αρνητική. Θα πρέπει λοιπόν στην πρότασή μας να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, διότι υπάρχουν κράτη-μέλη, υπάρχουν διάφορες περιοχές, ε, περιφέρειες, οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλά πώ να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρειαζόμαστε τι βέλτιστε πρακτικέ, διότι η αξία τη Ευρώπη είναι ακριβώ ότι μπορούμε να ανταλλάσσουμε τι βέλτιστε αυτέ πρακτικέ μεταξύ μα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό εάν θέλουμε να συμμετάσχει ε, και η βιομηχανία ε, η ε, Ευρώπη να έχει ηγετική θέση όσον αφορά την ενεργειακή τεχνολογία, διότι αυτό είναι κάτι που θα απασχολήσει όλον τον κόσμο στο μέλλον. Και τέλος, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με τα περιφερειακά ταμεία και το Ταμείο Σύγκληση για το πρόγραμμα αυτό, διότι όπω είπε ο συνάδελφο από τη Ρουμανία, φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προς τα νέα κράτη-μέλη, προ τι απόμακρε περιοχέ περιφέρειες και θα πρέπει όλα αυτά να αναφέρονται στα κριτήρια για τα νέα περιφερειακά ταμεία. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Ευχαριστώ. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κι εγώ κάτι. Εάν το θέμα σήμερα είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων, προφανώς η εμπειρία των κρατών μελών είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τι είδου εμπειρία έχει κάθε κράτο μέλο, σε ποιο τομέα, με τι αποτελέσματα, όπω είπε ο κύριο Πιπέρ νωρίτερα, όπου υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα, όπου λιγότερο καλά, με τι μέσα επετεύχθησαν. Όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε. Ο κύριος Πίπερ έχει πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν δώσατε επακριβείς απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις μου και θα πρέπει να επανέλθω. Για τους αδέρφους Γκίρεκ, Πρεζίνα και άλλους. Πάλι δεν δώσατε νομίζω τις σωστές απαντήσεις, γιατί στην απαντήση σας, εάν το βλέπω σωστά, εξισώνεται την εξοικονόμηση ενέργειας με την αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας. Με αποτέλεσμα το 1,5%. Εξοικονόμηση. Κάθε χρόνο και με στόχο δεσμευτικό για τους προμηθευτές ενέργειας στο ιδιωτικό νοικοκυριό. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω σε αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα δεν βλέπω καμιά δημιουργικότητα σε αυτές τις προτάσεις. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους, τα κράτη και τον ιδιώτη να αναπτύξουν νέες λύσεις, ε, να διδαχθούν ενδεχομένω και από αλλού, μεταφορά ε, τεχνογνωσίας, ε, κίνητρα, στόχοι. Δεν είναι δημιουργική λύση το να πείτε εξοικονόμηση σούτε με βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση. Πολλά ακόμα μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτόν. Επίσης και δυστυχώ δεν δώσατε απάντηση ικανοποιητική προ προς το μοντέλο των Primes. Ξέρω βεβαίω, είπατε κι εσεί ότι χρειάζεται βελτίωση το πρότυπο αυτό. Ε, λέτε όμως από την άλλη ότι ε, με βάση το επίπεδο ανάπτυξη του κάθε κράτους ε, του λέμε ότι θα πρέπει να βελτιώσει το επίπεδό του κατά 1,5%. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτοί που βρίσκονται στο υψηλότερο κλιμάκιο, στο υψηλότερο σκαλί της κλίμακας βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση. Γιατί κανείς δεν κοιτάει πώς θα γίνεται η μεταφορά το transfer δηλαδή από τον προς εκείνον που έχει το, τις χαμηλότερες επιδόσεις ή προς εκείνον που έχει τις καλύτερες επιδόσεις. Για όλους ισχύει ο όρος 1,5%. Δυστυχώς λοιπόν με πολύ περιορισμένη ε, δημιουργικότητα, πνεύμα παραγωγικό και φαντασία προχωράτε σε αυτά τα μέτρα. Πρέπει να κοιτάξουμε, η Σκανδιναβία, οι σκανδιναβικε χώρες, η Αυστρία θα υποχρεωθούν και εκείνε να φτάσουν σε 1,5% με τα ύψιστα ποσοστά που έχουν. Αυτό είναι μια ερώτηση μόνο. Αυτοί που έχουν ε, ανανεώσιμε πηγές σε τόσο καλή ε, ανάπτυξη θα πρέπει να παρουσιάσουν ε, περιορισμό στην χρήση των ανανεώσιμων κατά 1,5%. Και επίση έχω σπουδάσει γεωγραφία, χωροταξία χωροταξία περιβάλλοντος, ε, χωροταξία πόλεων. Και ξέρω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα εθνικό, μια προσέγγιση εθνική. Τώρα έρχεστε εσείς με τα ε, σχέδια αυτά τα οποία παρουσιάζετε να παρέμβετε μαζικά στην ε, κυριαρχία των κρατών και των κρατηδίων ή των περιφερειών και παραβιάζεται το άρθρο 94 το οποίο δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τέτοιου είδου ε, ε, παρέμβαση. Και έτσι θα ήθελα να δω αν έχετε κάποια άλλη νομική βάση που θα μπορούσε να αιτιολογήσει τέτοιου είδου μαζική παρέμβαση αρμοδιότητε των ε, κρατών μελών και των περιφερειών. Επίση, ω προ το κόστο που μπορεί να προκύψει για τον δημόσιο τομέα. Το 3% της υποχρέωσης για ανακαίνιση θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με το κράτος μέλος. Λαμβάνονται υπόψη στον προσδορισμό αυτού του 3% ότι εάν ο δημόσιο τομέας ή οι τοπικές περιφερειακές αρχές υποχρεωθούν να αγοράζουν μόνο ε, οικονομικά ως προς την χρήση ενέργειας ε, μηχανήματα ή εξοπλισμό μπορεί αυτό να, να οδηγήσει σε υψηλό κόστος, πολύ υψηλότερο μάλιστα σε κάποιον άλλο τομέα. Φερρυπίν, υποχρεούται ένας δήμος, μια κοινότητα να αγοράσει εκτυπωτή ε, οικονομικός προς την αξιοποίηση ενέργειας, αλλά αυτός έχει πολύ πιο ακριβό τόνερ για το μελάνι του. Αυτό λαμβάνεται υπόψη σαν κόστος ή κάτι αντίστοιχο που μπορεί να προκύψει στα συνέπεια. Λαμβάνονται αυτά όλα υπόψη στα σχέδιά σας ή μήπω τα ξεχάσατε κάπου. Σίσλι. Ευχαριστώ. Εδώ στα δεξιά σας, Πρόεδρε, δεν με βλέπετε και τόσο πολύ. Θα ήθελα για Θα ήθελα για την οδηγία αυτή να συζητήσουμε το θέμα της ε, υποχρέωσης για εξοικονόμηση κατά ένα 5% για τις επιχειρήσεις κάθε χρόνο και ως εκ τούτου εξοικονόμηση από κόστος για τον καταναλωτή, για τον πελάτη τους. Είπατε ότι ορισμένα κράτη, μέλη, έχουν μεγαλύτερο δυναμικό και άρα ίσως κάποια συστήματα δεσμευτικά που έχουν σταθεί σε κάποια κράτη-μέλη να μπορέσουν να εφαρμοστούν σε κάποια άλλα ή κάποια άλλα κράτη-μέλη ίσως να έχουν διαφορετική αντίληψη και ε, λύσεις για την εξοικονόμηση σε ενέργεια. Πώς λοιπόν θα μου δώσετε απάντηση στο θέμα των λοιπών εναλλακτικών που ενδεχομένω έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόψη με Φερρυπίν δημοσιονομικές λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Έχουν ληφθεί υπόψη τέτοιες προτάσεις, ιδέες και μια άλλη ερώτηση. Κάθε δεσμευτική διάταξη του νόμου απαιτεί και μια σχετική επένδυση. Πώς λοιπόν βλέπει την επίπτωση αυτών των δεσμευτικών διατάξεων ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έναντι ενδεχομένως άλλων προγραμμάτων, σχεδίων, έργων που αναπτύσσονται και είναι ενεξελίξει στα κράτη-μέλη και που ενδεχομένως θα αποστερηθούν από αυτούς τους πόρους. Επίσης μιλάτε για αυτό το 1,5% της ετήσιας εξοικονόμησης σε ενέργεια. Ταυτόχρονα εδώ εγγράφεται και το σύστημα της ανταλλαγής ε, εκπομπών, καυσε, ε, εκπομπών καυσέριων. Μπορείτε να μου δώσετε πιο πολλές εξηγήσει και πού βλέπετε συνέπεια στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριο Στούρμας. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι μιλάμε για ε, κυρώσεις. Κατά τη γνώμη μου, η οδηγία αυτή έχει να κάνει με ε, την μείωση της εξάρτησής μας από την ενέργεια, την ενίσχυση της παραγωγής, της ενέργειας και να ενισχύσουμε τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσον αφορά την ε, καινοτομία. Και ο κύριος Βέπερ ανέφερε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τον παγκόσμιο ανταγωνισμό ε, όσον αφορά την ε, ηγετική θέση για την ε, τεχνολογία αυτή. Η Κομισιόν στην μελέτη επιπτώσεων έχει εξετάσει αυτή την πτυχή, το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον ανταγωνισμό για την καινοτομία, διότι εάν παραμείνουμε στάσιμοι εδώ στην Ευρώπη και αυτός είναι κίνδυνος τώρα στην εποχή της κρίσης, σε έναν τομέα όπου ε, παλιά είχαμε την πρώτη θέση ε, απέναντι σε άλλες χώρες. Τώρα απειλούμαστε από χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χόν, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση. Ξέρω ότι πάντα ήταν δύσκολο να υπολογίσουμε την τελική χρήση ενέργειας, την τελική κατανάλωση ενέργειας. Ε, και υπήρχε ανησυχία ότι τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πολύπλοκα και δεν κάλυπταν τα πάντα. Και γι' αυτό ελήφθη η απόφαση ε, να πούμε και γι' αυτό έπρεπε να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο και καταλήξαμε πράγματι σε ένα ε, νούμερο όσον αφορά τον τελικό στόχο της ενέργειας μας ε, για το 2020. Εγώ νόμιζα πάντα ότι είναι εύκολο για την ε, Κομισιόν να υπολογίσει πόση ενέργεια καταναλώνει η Ευρώπη και μάλιστα κάθε κράτος μέλος, διότι υπάρχουν αυτές οι στατιστικές. Γιατί λοιπόν είναι τόσο δύσκολο να καταλήξουμε σε, μια, σε ένα στατιστικό νούμερο 20% ε, χαμηλότερο από την χρήση μας. Ε, νομίζω ότι ε, περιπλέκουμε τα πράγματα χωρίς λόγο. Η συνάδελφος Τόμσεν. Ναι, μερικές φορές όταν συζητάμε την απόδοση της ενέργειας, μου φαίνεται ότι περιπλέκουμε το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε και τα απλά ωφέλη. Εάν, για παράδειγμα, φέρουμε έναν εμπειρογνώμονα ε, εδώ στο Κοινοβούλιο, με μία μέρα μόνο θα μπορέσει να μας πει πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ε, το 20% της κατανάλωσης της ενέργειάς μας. Ε, αυτό είναι πολύ απλό και το κοινοβούλιο απλά πρέπει να επενδύσει, να ε, ε, εξοδεύσει την αμοιβή ενός ανθρώπου που θα έχει ένα μπλοκάκι και, ε, και, και μολύβι. Στη Δανία, για παράδειγμα, συνήθω δεν υπήρχαν θερμοστάτες στα σπίτια. Με την εγκατάσταση των θερμοστατών κάθε οικογένεια μπορούσε να αποφασίσει πόσο, πόσο ενέργεια θέλει να καταναλώσει. Ε, εξοικονόμησαμε πάρα πολλά χρήματα. Ε, στη Βαρσοβία, εάν ε, μειώσετε το θερμοστάτη κατά ένα βαθμό το, το χειμώνα μέσα στα σπίτια, μπορείτε να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα. Και αναφερθήκατε στις αγορές ΕΣΚΟ και θα ήθελα να γνωρίζω εάν η Κομισιόν εξετάζει την αγορά αυτή. Το ότι μία επιχείρηση πάει σε ένα νοσοκομείο και τους λέει ότι σας ε, προσφέρουμε ε, εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30% μας πληρώνετε και αν δεν έχετε καλύψει το, τα χρήματα αυτά μέσα σε δύο χρόνια, θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Αυτός είναι ένας τρόπος ε, να δείξει κανείς ότι ε, δεν στοιχίζει κάτι αυτή η επένδυση τελικά. Μήπως μπορείτε να μας ε, να εξετάσετε το θέμα αυτή, αυτού του τομέα. Ο συνάδελφος ε, Φανίστελ Ρόι. Για τα κίνητρα. Είναι πολύ απαγοητευτικό να διαπιστώνει κανείς ότι η Κομισιόν συνεχίζει το share management, τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων χωρίς να τα χρεξιοποιεί όμως. Ε, πρέπει να σταματήσει αυτή η παλιά μέθοδος των επιδοτήσεων, πρέπει να σκεφτούμε πιο μακροπρόθεσμα. Ε, δόθηκε το παράδειγμα των νοσοκομείων και να έχουμε πιο καινοτόμα και ε, μοντέλα και μέσα, οικονομικά μιλάμε. Στο νέο πλαίσιο λέει η Κομισιόν ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο, αλλά τελικά δεν θα πετύχουμε τίποτα, θα μειώσουμε την προσπάθεια άμα δεν αλλάξουν ουσιαστικά τα πράγματα. Δύο-τρει συνάδελφοι ήδη μίλησαν γι' αυτό. Και επειδή εγώ είμαι συγγητής για το νέο κανονισμό, αναρωτιέμαι Εάν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, ε, χωρίς μέσα διότι άμα τελικά εμείς ε, δεχθούμε περάσουμε λάθος μέσα και λάθος τρόπους εκτέλεσης δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα για να έχουμε πραγματική βελτίωση της κατάστασης πρέπει να έχουμε και μία αλλαγή νοτροπίας που θα τη συνοδεύει ο κύριος Χένεν ο κύριος ενέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Μου δημιουργεί μία σύγχυση όλη αυτή η συζήτηση. Εγώ δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Διότι άμα δεν δημιουργήσουμε κίνητρα δεν θα καταλήξουμε πουθενά η ενέργεια στοιχίζει όλο ένα και πιο ακριβά και στην παραγωγή και στους καταναλωτές. Άμα δεν συνειδητοποιήσουμε ότι πολλοί Ευρωπαίοι συμπολίτε δεν κατάφεραν να ζεσταθούν το χειμώνα διότι το κόστος της ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό για τα νοικοκυριά τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Και ένα, ε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Λοιπόν, κοινωνικές κατοικίες μιλάμε για ένα δημόσιο κτίριο, το οποίο όμως δεν θεωρείται πολλές φορές δημόσιο κτίριο γιατί θεωρείται κατοικία. Στις κοινωνικές κατοικίες ε, μένουν οι πιο φτωχοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να κάνουμε οικονομίες εγκαθιστώντας ε, νέους καυστήρες ε, φυσικού αερίου που καταναλώνουν 20% λιγότερο. Αλλά αυτό δεν αξίζει να το κάνουμε άμα δεν έχουμε μονώσεις στα παράθυρα. Διότι τότε δεν πετυχαίνουμε την οικονομία. Και εδώ χρειαζόμαστε βοήθεια, ενίσχυση για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικές οικονομίες. Δεν πρόκειται εδώ για εμπορικό τομέα όπου θα κερδίσει κάποιος επειδή ε, την οικονομία του φυσικού αερίου θα, θα την βάλει μετά στην τσέπη του. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους πιο φτωχούς καταναλωτές της Ευρώπης που θα έχουν ένα μικρότερο λογαριασμό που δεν θα γίνουν πλούσιοι Απλώς θα έχουν, θα, θα, θα, θα λίγο περισσότερη ευημερία να αφιερώσουν αυτή την εξοικονόμηση, αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσουν ε, για την τροφή τους ή οτιδήποτε άλλο. Τα κονδύλια λοιπόν πρέπει να χρησιμεύσουν για τη δημιουργία κινήτρων. Και οι, οι βουλευτές μπορούν να συζητούν και να διαπραγματεύονται με την Κομισιόν αλλά άμα δεν έχουμε κίνητρα τότε θα πρέπει να ψηφίσουμε καταναγκαστικά μέτρα. Διότι ο κόσμος δεν θέλει να κάνει οικονομίες. Και θα μπλεχτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα έχουμε δυσκολίες στην ίδια μας τη λειτουργία. Δεν βλέπω να στάει κανείς άλλο το λόγο, αλλά θα ήθελα και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Πάντοτε διστάζω να διατυπώνω ερωτήσεις που μπορεί να, κάνουν, να μας πάρουν χρόνο, αλλά ως προς την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί χωρίς να θεσπιστούν περαιτέρω μέτρα, όπως αναφέρει σελίδα 9, μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση στην ε, χρήση ενέργειας κατά 6% ε, δηλαδή εννοείται ότι μπορεί αυτή η ανταλλαγή εκπομπών αερίων να μην φέρει κανένα αποτέλεσμα ή δεν λαμβάνετε καθόλου υπόψη μελέτε σας. Επίσης, για τη στάση των κρατών μελών. Στη μελέτη επιπτώσεων λέτε ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν εισαγάγει μέτρα εξοικονόμηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, συγγνώμη. Ε, ρωτώ όμω, τα άλλα κράτη-μέλη τι στάση έχουν ακολουθήσει. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τα λοιπά κράτη-μέλη. Υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ αυτών διαφόρων μεθόδων ή συστημάτων που έχουν εισαγάγει τα διάφορα κράτη-μέλη. Η, η αλληλεπίδραση μεταξύ του συστήματος ανταλλαγών και των νέων συστημάτων ε, βελτίωση αποτελεσματικότητας έχει δώσει κάποια αποτελέσματα. Μας λέτε ότι υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση αλλά δεν έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχει κάτι να μας παρουσιάσετε. Μήπως τελικά θα έπρεπε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε ένα μέσον ε, για την επίδευση των στόχων, φέρει πίν την ανταλλαγή των ε, εκπομπών. Κοινωνικές επιπτώσεις, όπως αναφέρει και ο κύριος Σενά, τις ε, διερευνάτε, κοιτάτε τι γίνεται. Πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. Όταν λέτε ότι τα παρεπόμενα, οι παρεπόμενες δαπάνες μπορεί να μειωθούν στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, τι συνέπειες βλέπετε μπορεί να υπάρξουν μέτρα εξοικονόμησης, μάλλον εξυγίανσης της ενεργειακής χρήσης. Γιατί, παραδείγματι, στην πατρίδα μου αναφέρονται πολύ συχνά φόβοι ότι ένα σύστημα με την ανακαίνιση ε, κατοικιών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ενοικίων κατά 70% πράγμα το οποίο δεν θα προξενούσε ένα άλλο σύστημα, μια άλλη μέθοδος ανακαίνησης. σε αυτό έχετε κάνει κάποιες μελέτες και ο κύριος ε, Βέμπερ που μίλησε για τα FEE δίκτυα. Η εξοικονόμηση ενεργησίας ανάλογα με το μοντέλο που ακολουθείτε είναι στο 0 ε, ή μέχρι το 10%. Εάν δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό γίνεται εξοικονόμηση, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την χρήση αυτών των εφιών δικτύων. Έχω και άλλες ερωτήσεις βέβαια, αλλά μπορώ να περιμένω. Το θέμα είναι να διευκρινίσουμε ορισμένα ζητήματα με τις ερωτήσεις μας, ορισμένες λεπτομέρειες. Ο κύριος Πίπερ βλέπω ότι θα πάλι το λόγο. Και μετά στο βαθμό βέβαια που μπορείτε θα μας δώσετε τις απαντήσεις. Κύριε Σπίπερ, εδώ πολλοί συνάδελφοι παραπέμπουν στα ερωτικά ταμεία και λένε ότι θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε περισσότερο για τη βελτίωση, την επίτευξη μάλλον των στόχων της αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας. Μία περιφέρεια η οποία έχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, μεγάλο προσδόκιμο ανάπτυξης ε, περιμένει ότι θα έχει καλή ε, και μεταφορά ενέργειας μπορεί να επενδύσει και εξοικονόμηση μεταφορά τεχνογνωσίας μπορεί να επενδύσει και υποδομές ε, και εξοικονόμηση ενέργειας. Φερπίν μια περιφέρεια ανεπτυγμένη σε ένα μικρό κρατοσμένος και ταυτόχρονα υποχρεούται να μειώσει κατά 1,5% κάθε χρόνο το την ε, κατανάλωση ενέργειας. Τι είδους προοπτικές ανάπτυξης μπορεί να έχει μια τέτοια περιοχή, μια τέτοια περιφέρεια. Και επίσης στα διαρθρωτικά ταμεία στα ΕΦΗ, e e δίκτυα θα πρέπει να επενδύουμε μάλλον παρά σε ε, άλλες παραγωγικές ε, μονάδες γιατί καταλαβαίνω βεβαίως ότι είναι πολύ καλή η λύση της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά το 20% των διαδοτικών ταμείων θα πρέπει να αφοσιωθεί μόνο στον τομέα αυτών, πιστεύω θα αποτελεί μια πολύ εσφαλμένη επιλογή και πολύ κακό ε, βήμα σε σχέση με τους στόχους της ανάπτυξης. Κύριε Χάντσεν για να απαντήσω. Ευχαριστώ και πάλι. Η κυρία Τόμσεν ανέφερε ότι η Δανία ως κράτος μέλος ε, στήριξε την ιδέα του δεσμευτικού στόχου και μας ρωτάει γιατί δεν ε, ακολουθήσαμε αυτόν τον δρόμο. Η Δανία ήταν η μόνη χώρα που ήθελε δεσμευτικούς στόχους. Και γι' αυτό, πέρα από τη συζήτηση για το ωφέλη της μίας ή της άλλης προσέγγισης, ε, λάβαμε ένα πολύ σαφέ ε, μήνυμα από τη μία από το Κοινοβούλιο, αλλά από το Συμβούλιο λάβαμε ακριβώ το αντίθετο μήνυμα και γι' αυτό υποβάλαμε μία πρόταση ε, σε δύο στάδια, ε, στην οποία το πρώτο στάδιο είναι δεσμευτικά μέτρα, τα οποία πιστεύουμε ότι θα μας... μη δεσμευτικά μέτρα, τα οποία πιστεύουμε ότι θα μας Συγγνώμη, το, στάδιο 1 για τα δεσμευτικά μέτρα που πιστεύουμε ότι θα ε, μας βοηθήσουν να πετύχουμε τον στόχο μας ε, και αν δεν πετύχουμε αυτό, τότε θα προχωρήσουμε στο στάδιο 2 με δεσμευτικούς στόχους. Ε, ε, υπάρχουν ωφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν από τους δεσμευτικούς στόχους. Υπάρχουν όμως ε, και άλλοι τρόποι να πετύχουμε αυτά, όπως για παράδειγμα ο οικολογικός σχεδιασμός υιοθετώντας ε, φιλόδοξα ελάχιστα πρότυπα ε, ε, και συνδέοντάς τα με τα πρότυπα για τις μετρήσεις θα πετύχουμε πολλά. Διάφοροι και οι Κινέζοι έρχονται και μας ρωτάνε πώς τα καταφέρνουμε όλα αυτά. Ε, γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά ότι πρέπει να πετύχουμε τους στόχους μας αυτούς. Όσον αφορά το πολιετές ε, πλαίσιο που αναφέρατε και εσείς και άλλοι, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πω ποια θα είναι η πρόταση της Επιτροπής. Ε, τον επόμενο μήνα θα υποβάλουμε πρόταση, αλλά γνωρίζετε από την ανακοίνωση του Ιουνίου ότι όπως είπε και ο κύριος Πίπερ υπάρχει Υπάρχουν σημαντικέ δυνατότητε για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ε, θέλουμε να υποβάλουμε μια πρόταση που να ενσωματώνει την προσέγγιση αυτή και είναι σαφέ από την συζήτηση που είχαμε ότι αυτό θα συζητηθεί σε, πολλά, σε πολλού χώρου του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Πίπερ ε, ρώτησε τι γίνεται με τις προσπάθειες να μάθουμε από τις ε, βέλτιστες πρακτικές των διαφόρων κρατών μελών. Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας αυτή. Ένας ε, λόγος ε, που ε, πολλά πράγματα δεν γίνονται είναι ότι είναι πολύπλοκα και απαιτούν ειδικέ γνώσεις. Τα στηρίζουμε αυτά με συντονισμένες δράσεις, με διάφορα προγράμματα όπου συμμετέχουν άνθρωποι από διάφορα κράτη-μέλη με σκοπό την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και ε, μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι οι ε, γερμανικοί επιρογνώμονες συμμετέχουν επίσης στα προγράμματα αυτά. Θέλουμε οι επιρογνώμονες από διάφορους τομείς να μοιραστούν με άλλους τις γνώσεις τους. συμφωνώ με αυτό που είπατε, απλά δεν αποτελεί μέρος της συγκεκριμένη πρότασης. Όσον αφορά το 1,5% θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται για περικοπή κατά 1,5%. Δεν ζητάμε μείωση 1,5% το χρόνο στην κατανάλωση. Αυτό που ζητάμε ή που προτείνουμε ε, είναι οι προμηθευτές ενέργειας να δείχνουν ότι έχουν κάτι το οποίο να ε, εξοικονομεί ε, κάτι το οποίο να αντιστοιχεί στο 1,5% των πωλήσεων της προηγούμενης χρονιάς. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση πουλάει 100 το, το έτος Χ, το επόμενο έτος ε, θα πρέπει, για παράδειγμα, να έχει εγκαταστήσει μονοτικά παράθυρα ή νέους καυστήρες, ε, ώστε ε, να υπάρχει εξοικονόμηση που να αντιστοιχεί στο 1,5. Μπορεί όμως, αν υπάρχει μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας, να υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης, δηλαδή στο 102 να βρίσκεται η κατανάλωση την επόμενη χρονιά, αλλά χωρίς τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων να έφτανε το 103 ε, και μισό. Χώρες ε, με πολύ ανανεώσιμη ενέργεια θα πρέπει και αυτές να εξοικονομήσουν. Αναφέρατε την Σκανδιναβία και την Αυστρία. Και εμεί ε, το πιστεύουμε αυτό, η βιομάζα που είναι ο πόρος που χρησιμοποιούν ε, ε, είναι περιορισμένο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερη βιομάζα για να πετύχουμε τους ε, ενεργειακού μα στόχους. Θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικούς καυστήρες για βιομάζας όπως απαιτούνται και αποτελεσματικοί καυστήρες για τον άνθρακα. Δεν οδηγεί σε εξαίρεση δηλαδή από τους στόχους εάν κάποιος έχει υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όσον αφορά το θέμα της επικουρικότητας που αναφέρατε, Η πρόταση αυτή έχει ως νομική βάση το άρθρο 194 της συνθήκης, το οποίο είναι το νέο ε, άρθρο για την ενέργεια. Ο στόχος του είναι ενεργειακός. Και κατά τη δική μας εκτίμηση είναι απόλυτα σωστό ο στόχος αυτός να επιτευχθεί ε, με διάφορα μέσα και ένα από αυτά, όχι το πιο σημαντικό, αλλά ένα από τα στοιχεία είναι κάποιες απαιτήσει που έχουν να κάνουν με, με την ε, χωροταξία. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα αυτό να είναι μέρος της ε, συνολικής ε, πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 194. Εάν ήταν μια καθαρά περιβαλλοντική πρόταση, και στηριζόταν στη νομική βάση του άρθρου 192, τότε τα στοιχεία αυτά θα έπρεπε να υιοθετηθούν με ομοφωνία στο Συμβούλιο, αλλά δεν είναι περιβαλλοντική η πρόταση αυτή, είναι ενεργειακή και σίγουρα θα πρέπει να υποφεληθούμε από τις νέες αρμοδιότητες στον χώρο της ενέργειας που μας ε, δίνει η συνθήκη. Γι' αυτό δεν ε, προκύπτει πρόβλημα. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά αν θέλετε, αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε εξετάσει και είμαστε βέβαιοι όσον αφορά την ε, εκτίμησή μας. Όσον αφορά το επιπλέον κόστος για τον δημόσιο τομέα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι μιλάμε για μείωση του κόστους ε, κατά την ε, χρήση ε, του εξοπλισμού αυτού. Αν αγοράσει κανείς δηλαδή καλύτερο εκτυπωτή, ο οποίος είναι πιο ακριβώς, είναι πιο αποδοτικός, θα χρησιμοποιεί κάθε, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, θα, θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και έτσι το συνολικό κόστος ε, στο δημόσιο τομέα ε, θα μειωθεί σημαντικά. Ε, πρόβλημα στο δημόσιο τομέα είναι ότι οι αποφάσεις συχνά λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση το κόστος. Ποια είναι δηλαδή η φθηνότερη συσκευή που μπορεί να αγοράσει κανείς χωρίς να εξετάζει το κόστος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Γι' αυτό ζητάμε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη και τη διάρκεια ζωής του, της συγκεκριμένη μηχανή. ρωτήθηκε επίσης αν εξετάζουμε εναλλακτικέ λύσεις σε σχέση με την, ε, με, την απέτηση για μείωση κατά 1,5%. Ε, μιλώ για εναλλακτικέ λύσει στα υποχρεωτικά ε, προγράμματα. Ναι, ακριβώ αυτό εννοούσα, λέει ο μιλητή. Όπω ανέφερε ο κύριο Τούρμε, ε, το άρθρο 6, παράγραφο 9, ε, αφήνει χώρο ε, στα κράτη-μέλη, επιτρέπει κάποιο περιθώριο στα κράτη-μέλη για να έχουν εναλλακτικέ ε, προσεγγίσεις. Ε, δεν αναφέρεται... Δεν αναπτύσσεται αναλυτικά αυτό. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου μπορούν να οδηγήσουν σε προσθήκη περισσότερων λεπτομεριών, όπως και η συζητήσεις στο Κοινοβούλιο μπορεί να οδηγήσουν ε, σε πιο αναλυτική διατύπωση. Ε, όποιος ε, λοιπόν διαβάσει το άρθρο 6 παράγραφος 9 μπορεί να θέλει μια πιο αναλυτική εκτίμηση. Πάντως αυτό που είπαμε στο Συμβούλιο και που λέμε και σε εσά είναι ότι ευχαρίστω θα υποβάλουμε τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση υποβληθεί. Η ε, μελέτη επιπτώσεων ε, εξετάζει και το διοικητικό κόστος ε, και τις άλλες σχετικές δαπάνες. Ναι, συμπεριλαμβάνονται. Όσον αφορά την επιπτώ... τις επιπτώσεις στη χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων, όπως σας είπα, στόχος είναι να, να μπορούν να διατεθούν περισσότερα χρήματα για άλλα προγράμματα. το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα ήταν λογικά να γίνουν, τα οποία όμως δεν ε, γίνονται. Για παράδειγμα, ε, ξέρουμε ότι πολλοί κόσμος ε, μένει σε σπίτια που δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα ε, ή επίση ξέρουμε ότι παρότι τελικά οδηγούν σε εξοικονόμηση τα μέτρα αυτά, το αρχικό κόστο είναι πολύ μεγάλο. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε το κόστος αυτό. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να κάνει παράλογα πράγματα. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να κάνει τα πράγματα που θα οδηγήσουν τελικά σε εξοικονόμηση. Ε, όλα αυτά ε, είναι συμβατά με το πρόγραμμα ε, εμπορίας εκπομπών. ναι, κατά τη γνώμη μας είναι. θα πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις ε, στο ε, πρόγραμμα εμπορίας εκπομπών, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει ασύμβατότητα. Πιστεύουμε ότι είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους αυτά τα δύο. Ο κύριος ε, Τούρμες μίλησε για τις επιπτώσεις στην καινοτομία. Αυτό μόνο σε περιορισμένο βαθμό λαμβάνεται υπόψη εδώ πέρα. Το πρότυπο που εξετάσαμε αναγνωρίζει εν μέρη ότι εάν αναπτυχθεί αγορά για μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή ε, προϊόν, ε, τότε θα ε, μειωθεί το κόστος, αλλά δεν εξετάζουμε αναλυτικά μεμονωμένα κάθε υπηρεσία ή κάθε προϊόν. Αυτές οι εκτιμήσεις δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί στην μελέτη μας. Η κυρία Χολ ρώτησε αν ε, ο συνολικός στόχος για την Ευρώπη το 2020 ε, είναι ενέργεια που να αντιστοιχεί σε 1.374.000 ε, τόνους πετρελαίου, γιατί δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε και τον στόχο μας. Η απόφασή μας δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα τεχνικό πρόβλημα. Θέλουμε να επιλέξουμε τον σωστό δρόμο να προχωρήσουμε. Τούτο λεχθέντος Υπάρχουν διάφοροι κανόνες ε, που θα μπορούσε κανείς ε, να ε, επινοήσει για να μοιράσει αυτό το νούμερο που σας έδωσα και μπορούν να γίνουν διάφορες επικρίσεις για τους κανόνες αυτούς σχετικά με το πώς κοιτάνε τις δυνατότητες, τους περιορισμούς των, των διαφορών κρατών μελών. Εάν είχαμε υποβάλει μια τέτοια πρόταση, σίγουρα δεν θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να έχει γίνει εύκολα και γρήγορα. Κυρία Τόμσεν, ε, από την απάντηση προς την κυρία Γιώργα Στελιά ε, θα καταλάβατε ότι συμφωνώ μαζί σας ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν ε, τα οποία απαιτούν ένας εμπειρογνώμου να κάνει ένα γύρο με ένα μπλοκάκι και ένα μολύβι. Ναι, εξετάζουμε την αγορά. Σκό, θα σας στείλω τους ε, ηλεκτρονικούς συνδέσμους ε, για κάποιες μελέτες που ήδη έχουμε κάνει. Ε, μεγάλο μέρος των βέλτιστων πρακτικών προέρχονται από την Γερμανία. Είδαμε όμως και κάποιες πολύ καλές πρακτικές από τη Δανία, τις οποίες θα θέλαμε να διαθέσουμε ευρύτερα. Κύριε Φανίστελ Ρόι, ναι, συμμερίζομαι τη δυσαρέσκειά σας. Υπήρχε πρόβλεψη στα διαρθρωτικά ταμεία για την ενεργειακή απόδοση στην ε, παρούσα προγραμματική περίοδο δεν ε, ε, έχει χρησιμοποιηθεί, κυρίως επειδή χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεση τροποποίηση των κανόνων. Δεν θα έλεγα ότι είναι λάθος η χρήση των διαθροτικών ταμείων, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε πιο, πιο καλές προσεγγίσεις και Έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε αυτό σε μικρή κλίμακα, για παράδειγμα με το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης. Ε, συνεργαζόμαστε με τράπεζες ε, για να καταλάβουν καλύτερα την ε, αγορά ενεργειακής απόδοσης. Έχουμε το πρόγραμμα Ελένα, το οποίο συνεργάζεται με τοπικές αρχές για να καταλάβουν καλύτερα τις τράπεζες για να μπορούν να συνδυάζονται προγράμματα ενεργειακή απόδοση. Ε, ελπίζουμε όλα αυτά να μπορέσουν τελικά να ενσωματωθούν στα διαστατικά ταμεία και ελπίζουμε ότι και τα κράτη-μέλη θα το κάνουν αυτό, ε, διότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο κύριο Ανά μίλησε για τις επιπτώσεις ε, στις κατοικίες και ιδιαίτερα τις κοινωνικές κατοικίες. Όπως θα γνωρίζετε, οι κοινωνικές κατοικίες συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 4 ε, σχετικά με την ε, βελτίωση ε, κατά 3% των κατοικιών κάθε χρόνο. Τουλάχιστον μιλάμε για τα μεγάλα συγκροτήματα κοινωνικών κατοικιών, διότι τα μέτρα αυτά περιορίζονται στα μεγάλα κτίρια. Ο κύριος Πίπερ αναφέρθηκε στο κόστος για τους ενίκους. Ναι, βλέπουμε ότι όσοι μένουν σε κοινωνικές κατοικίες θα υποφεληθούν από πιο ε, ε, ε αποδοτικά ενεργειακά κτίρια, για παράδειγμα ε, σε σχέση με το αν δεν έχουν θερμοστάτες. Πώς μπορεί να διασφαλίσουμε, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας δεν, δεν θα είναι εις βάρος των ανθρώπων με χαμηλότερο εισόδημα θα υπάρχει επιδότηση για το αρχικό στάδιο, όχι όμως για το σύνολο της ε, δαπάνης. Ε, στην περίπτωση αυτή, ε, όποιος δεν έχει χρήματα, δεν θα μπορέσει να συμπληρώσει το υπόλοιπο, αλλά θα, παρόλα αυτά θα δει τα ωφέλη από την μελλοντική εξοικονόμηση. Και Θέλουμε τα κράτη-μέλη να φροντίσουν, ε, να διαχειριστούν το πρόγραμμα αυτό έτσι, ώστε να μην αποφεληθούν ε, μόνο οι πιο ευκατάστατοι, αλλά και ε, οι άνθρωποι με χαμηλότερο εισόδημα. Επίσης, κύριε Ροελ, το πρόγραμμα εμπορίες εκπομπών, ενώ έχει παρουσιάσει σημαντικά ωφέλη, δεν έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη αλλαγή κατεύθυνση ε, όσον αφορά τις ε, πηγές ενέργειας. Και αναρωτιόμαστε αν ε, αυτό θα συνεχίσει να ισχύει και κατά την τρίτο περίοδο του προγράμματος αυτού, εάν δεν δούμε ούτε εδώ αλλαγή κατεύθυνση, ε, τότε μπορεί να επανέλθουμε με συγκεκριμένε απαιτήσει για τον τομέα αυτόν. Είναι δυνατόν λοιπόν το σύστημα εμπορίας εκπομπών ε, να ε, εξαντλήσει τις δυνατότητες αυτές, αλλά τα στοιχεία που έχουμε σήμερα μας δείχνουν ότι δεν έχει γίνει αυτό στο βαθμό που επιθυμούσαμε. Το δανέζικο, γαλλικό, ε, ε, βρετανικό και φλαμαντικό σύστημα έχουν ε, μεγάλες αλλαγές μεταξύ τους και η κυρία Φόρντ αναφέρθηκε σε αυτό νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Όλα λειτουργούν, όλα έχουν οδηγήσει σε εξοικονόμηση. Υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες ομοιότητες, για παράδειγμα, παρότι κάποια από τα προγράμματα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να πετύχουν εξοικονόμηση όχι μόνο από τους δικούς τους πελάτες αλλά και από πελάτες άλλων, ε, στην πραγματικότητα η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται μεταξύ των πελατών ε, της ίδιας της επιχείρησης, ε, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον εξοικονομήσεις εδώ πέρα. Θα μπορούσα να στείλω στους βοηθούς σας τις σχετικές μας εκτιμήσεις. Ανέφερα ήδη τις κοινωνικές επιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε αρνητικές κοινωνικές ε, επιπτώσεις ε, και μάλιστα το βρετανικό ε, πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα καλής πρακτική. Όσον αφορά τι κοινωνικέ κατοικίε και το τι θα γίνει με το 3%, αυτό πράγματι συνδέεται με το ερώτημα πώς θα, στηρί... μοιράσουμε το κόστος και τα ωφέλη μεταξύ των ενίκων. Οι ευφυείς μετρητές όπως είπατε, προσφέρουν ε, περιορισμένα ε, ωφέλη. Αν όμως ε, έχουμε πιο συχνή τιμολόγηση, τότε θα δούμε μεγαλύτερα ωφέλη, διότι έτσι αντικατοπτρίζονται καλύτερα ε, οι εξοικονομήσει. Κύριε Πίπερ, συμφωνώ ότι τα διαφορετικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, για να δούμε τεχνική και τεχνολογική πρόοδο. Όπως είπαμε, η, απόδοση, η ενεργειακή απόδοση βοηθάει σε αυτό, αλλά ε, δεν μιλάμε για 100% ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει να δούμε την όλη ισορροπία εδώ. Και ελπίζω έτσι ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Έχω ζητήσει ακόμα συναδελφοί το λόγο. κυρία Τόμψεν, για το ερώτημά μου, εάν χώρες οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει σε μείωση υποχρεούνται να συνεχίσουν να μειώνουν. Δηλαδή, βασικά, τι δυναμικό έχουμε μέσα στην αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Πρόσφατα, η, ε, το επιμελητήριο, της το επιμελητήριο των μηχανικών Δανίας ε, έδωσε κάποιες ενδείξεις και συμβουλές για το πώς θα, κάνουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας και θα μπορούσαμε να τους προσκαλέσουμε εδώ σε μια ακρόαση για να μας δώσουν τις συμβουλές τους. Γκλάντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή κύριε Χάντσεν. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από τις ε, τελευταίες απαντήσεις ε, με ακόμα δύο ερωτηματικά. μία επιχείρηση προμήθειας ενέργειας, όχι παραγωγής, προμήθειας μόνο με την οποία έχω συνομιλήσει πρόσφατα, μου εξήγησε τι είδους επιχειρηματικά μοντέλα μπορεί να, έχει, ε, να εφαρμόσει για βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση ενέργεια. Πλην όμως, ένα νοικοκυριό το οποίο δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δαπάνη δεν είναι και σε θέση να εισαγάγει ένα εξοπλισμό όπως σύγχρονο σύστημα θέρμανσης με λέβητα οικονομικό κτλ. Και άρα δεν μπορεί να ανθέξει το σχετικό κόστος. Άρα θα πρέπει ο προμηθευτής αυτός να του καλύψει τη σχετική δαπάνη με μια δέσμευση μακροπρόθεσμη εκ μέρους του ε, καταναλωτή για ε, συμβόλαιο ε, προμήθειας φυσικού αερίου φερρυπίν από το συγκεκριμένο προμηθευτή. Αλλά αυτό δεν προβλέπεται. Επίσης το smart battering ή το smart grid, τα FEE δίκτυα, θα πρέπει να είναι τέτοια η ικανότητά τους να δώσουν ε, καταμέτρηση κόστους και κατανάλωσης που να επιτρέπει και στον, στη ρυθμιστική αρχή να ε, τροποποιήσει αντίστοιχα τα τέλη κατανάλωσης ενέργεια. Πράγμα το οποίο στη Γερμανία τουλάχιστον δεν ισχύει ακόμη. Ο κύριο Τουρμέ δεν θέλω ευχαριστώ. Χωρί μικρόφωνο. Κύριο Στουρμέ. νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση πιστεύω θα πρέπει να πούμε το εξωτερικό. θα πρέπει να χάσουμε την ε, γενική εικόνα που είναι η ανεξαρτησία από τις ενεργειακές ή η μείωση της εξάρτησης από τις ενεργειακές ε, πηγές ή ε, κυρίως αυτές που βρίσκονται εκτός Ευρώπης αλλά ταυτόχρονα και αναζήτηση πιο καινοτόμων ε, μέσων μια υποχρέωση φερρυπίν καινοτομία που εισήχθηκε στη Γερμανία, στην Γαλλία, την Ιταλία, το Ρωμένο Βασίλειο αποτελεί μια λύση την οποία τουλάχιστον οι ειδικοί όταν ε, μας ε, εξηγούν τις θέσεις τους, βλέπουν ότι μπορεί να εξοικονομήσει δαπάνες από δαπάνες και να δώσει αποτελέσματα πολύ καλύτερα από ότι ε, οι επενδύσεις οι κρατικές μέχρι τώρα. Στη Γερμανία, Φερρυπίν, αυτή η πρώτη ιδέα της γερμανικής κυβέρνησης για μείωση η έκπτωση φόρου κατά, περικοπή μάλλον φόρου κατά 1,5 δισεκατομμύριο Φαίνεται ότι τώρα βρίσκεται σε παιδό ε, μπλοκαρισμένη, δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί δεν εγκρίνεται από τον Bundestag. Άρα ίσως θα πρέπει να δούμε εάν μια τέτοια υποχρέωση εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί ακόμα και για τη Γερμανία να φέρει ε, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βέβαια αυτό ακόμα δεν έχει κριθεί, θα το δούμε στο μέλλον. Το θέμα είναι πώς τα παλαιά επιχειρηματικά μοντέλα, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, η παλαιά βιομηχανική παραγωγή με την σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή μπορούν να συνεργαστούν σε αυτό το τομέα. Και εμείς ως υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής στον ευρωπαϊκό κλάδο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε προτάσεις και αυτό ίσως να ε, περιλάβω εγώ σε μια πρόταση για την ε, προσφορά και ζήτηση ή μάλλον ανταπόκριση στη ζήτηση με στόχο να δώσω περισσότερα κίνητρα στην ε, παραγωγή την ευρωπαϊκή. Αλλά επαναλαμβάνω δεν πρέπει να ξεχνάμε ποια είναι η γενική εικόνα ότι έχουμε να εξοικονομήσουμε αυτά τα 300 κάτι δισεκατομμύρια τόνους του πετρελαίου Και εάν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι στον τομέα, θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες και περικοπές των άλλων. Ευχαριστώ. Εάν θέλετε για τι δύο παρατηρήσει να προσθέσετε κάτι, εσείς παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ τα σχόλια των, ε, της κυρίας Τόμψεν και του κύριου Τουρμές δεν ήταν ερωτήσεις για μένα, αλλά δεν έχω να σχολιάσω. Για τον κύριο Γκλάντε όμως, το ερώτημα για τα εφή δίκτυα δεν είναι ακριβώς αντικείμενο της δικής μας προτάσεως, αλλά είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί. Η ιδέα του Λέβητα είναι μια ιδέα ε, που πρέπει να προωθηθεί, δηλαδή να βρούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι, οι πιο οικονομικοί και οι πιο αποτελεσματικοί, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές των ε, Λεβίτων, ειδικά για τους πιο αποτελεσματικούς στην ε, χρήση ενέργειας. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ρόιλε. Ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε τόσο χρόνο στη θέσή μα ε, σήμερα. Συνήθω έχουμε πολύ περιμένη ημερήσια διάταξη. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν λεπτομερέστατα να δούμε τα θέματα αυτά. Φυσικά, εάν θέλουν επιμέρου ζητήματα να διατυπώσουν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, οι συνάδελφοι γραπτός ε, προς τη γραμματεία παρακαλώ για να τα διαβιβάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάλι οι αποφάσεις, οι απαντήσεις θα ε, διατεθούν και στους συναδέλφους. Η μελέτη αξιολόγηση θα εξεταστεί εσωτερικά στην Επιτροπή μας την επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ολοκληρώσαμε το τρίτο. Κυρία Χάντσελ, σας ευχαριστώ πολύ και χαίρετε. Και περνάμε κυρίες και κύριοι. Προχωράμε με θάρρος και παρησία. Για να δούμε. Κυρίε και κύριοι, σημείο 4, ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου του Συμβουλού την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, το ανοιχτό διαδίκτυο και η δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη. Ε, βλέπω ότι αδειάζει η αίθουσα, τάχιστα, όπως είχαμε προβλέψει. Έχουμε καταθέσει προφορική ερώτηση και πρώτο σχέδιο ψηφίσματος για την πρόταση αυτή. Το έχουμε επεξεργαστεί. Το ψήφισμα αυτό δεν θα σας καθυστερήσω. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο με μια πιο ταχεία διαδικασία. Αυτό είναι και το σχέδιό μας λίγο. Εάν θέλετε όμως να δώσω σύντομα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μας πει δύο λόγια. Είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς εκ της Επιτροπής σε θέση, Μπρίνκαλτ, ποιος είναι, για να μας εξηγήσει εδώ τα... Δύο-τρία λόγια μόνο σας παρακαλώ. Η σειρά σας. Και μετά η κυρία Ματουρέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ρόιλ που μας έδωσε το λόγο. Μετά την έγκριση της ανακοίνωσης την τελευταία περασμένη άνοιξη, τώρα έχουμε μια συζήτηση για την καταγραφή της κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα περιμένουμε και την εφαρμογή του πακέτου των τηλεπικοινωνιών του 2009 από τα κράτη-μέλη, γιατί δεν το έχουν εφαρμόσει όλα τα κράτη-μέλη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και επίσης εξετάζουμε και τις μελέτες των οικονομικών επιπτώσεων. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαντουρέλ παρακαλώ τότε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα. Εμείς συμφωνούμε με το κείμενο της ερώτησης και για την ευστοχία της και για τους λόγους που αναφέρονται και στην ερώτηση την ίδια. Τώρα για το ψήφισμα η συγκήτριά μας που δυστυχώς σήμερα απουσιάζει και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της μου έστειλε ορισμένα σχόλια τα οποία θα σας πω πολύ σύντομα. Πρώτο, σχετικά με δύο εκτιμώντας. Θεωρούμε ότι το δέλτα, το D, πρέπει να είναι σαφέστερο ως προς την αρμοδιότητες του ΕΡΕΚ Τα international scale θέλουμε να τα αλλάξουμε με, με τον όρο cross border scale και για τα άρθρα έχουμε μερικά σχόλια. Για το 2 θεωρούμε ότι δεν πρέπει να είναι τόσο κατηγορηματικό διότι η ανάλυση στην οποία αναφέρεται είναι κάτι που αμφισβήτησε τόσο η βιομηχανία όσο και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Με το 7 δεν συμφωνούμε με την έκφραση μία λογική εργασία και θα θέλαμε να προσθέσουμε και τέσσερα σημεία ως εξής. Πρώτον, να διατηρηθεί ως κανόνας το best effort internet, η βέλτιστη προσπάθεια διαδικτύου, Με μετά δεύτερο σημείο για το EPTV, ε, τρίτο ότι εγγυόμαστε την δυνατότητα καινοτομίας χωρίς εμπόδια και τέταρτο ότι η αγορά ε, διαδικτύου έχει δύο πλευρές. Αφενός τους διαχειριστές και μετά τις επιχειρήσεις ε, τηλεπικοινωνίας. Θέλουμε την ουδετερότητα του δικτύου επίσης και θέλουμε να έχουμε και τον όρο device neutrality. Στην περίπτωση δηλαδή των ε, smartphones όπου δεν μπορούμε να ε, παίρνουμε λογισμικό και δεν έχουμε περιθώριο δηλαδή, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Βανίστερο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα κι εγώ. Εμείς βρισκόμαστε σε μια φάση όπου είναι καλό να έχουμε καλές πληροφορίες και να έχουμε υπόψη μας και ποιες είναι οι αρχές που κρύβονται στη βάση όλων αυτών. Εγώ συμφωνώ με το κείμενο, όμως ε, μερικά άλλα στοιχεία πρέπει να τα τονίσουμε ή να τα ενισχύσουμε. Είναι ενδιαφέρον να να δούμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων σε ορισμένα κράτη-μέλη. Διότι σε ορισμένα κράτη-μέλη έχουμε νομοθεσία σχετικά. Πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της. Δεν μπορούμε όμως να επιτρέπουμε ένας διανομέας να συμπεριφέρεται σε μια χώρα προς έναν καταναλωτή διαφορετικά από ό,τι σε μια άλλη χώρα διότι τα πάντα είναι διασυνοριακά. Πρέπει να έχουμε κατά συνέπεια μια νομοθεσία που δεν θα επιτρέπει μόνο περισσότερη χρηματοδότηση για καλύτερη πρόσβαση στο δίκτυο αυτό. Συμβαίνει σε πολλά κράτη-μέλη ήδη θα χρειαζόντουσαν ίσως μελέτες και να λάβουμε μία απόφαση αργότερα. Υπάρχουν μοντέλα τα οποία πραγματικά είναι καλά. Υπάρχουν επιχειρήσεις, εταιρείε οι οποίες μπορούν να προσφέρουν καλές τιμές διότι επένδυσαν στα δίκτυα οπότε σήμερα μπορούν να ε, ανασύρουν και τα πλεονεκτήματα. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να έχουμε, να σκεφτούμε μάλλον, ότι πολλές χώρες συζητάνε ακόμα το τι είδους νομοθεσία θέλουν να εφαρμόσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση. Να δούμε τι επιπτώσεις είχαμε στις χώρες όπου υπάρχει ήδη νομοθεσία ή όπου συζητείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι και εξαντλήθηκαν τώρα οι παρεμβάσεις. Θα σας παρακαλέσω, εάν έχετε κάτι συγκεκριμένο για προτάσεις, να μας το δώσετε γραπτός και θα το επεξεργαστούμε ακόμη το κείμενο και φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε και κάποιες προτάσεις από τις ε, άλλες επιτροπές των οικονομικών, της ιστορικής αγοράς μάλλον κτλ. 20 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία για τις τροπολογίες 12, ε, στα αγγλικά, παρακαλώ για το ψήφισμα. Αλλά χωριστά τώρα το ζήτημα της προφορικής ερώτησης. Ως προς τη διατύπωση της ερώτησης δεν βλέπω να υπάρχουν επιφυλάξεις, ε, μπορούμε να τη δώσουμε, να την καταθέσουμε δηλαδή. Άρα, κλείνει το θέμα της ερώτησης για δε το ψήφισμα ή προτάσεις όπως τις ορίζει το χρονοδιάγραμμα 20 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι και εκεί κλείνουμε και την προθεσμία για την κατάθεση. Άλλες επιφυλάξεις υπάρχουν όχι. Πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Προχωρούμε ταχύτατα και σας ευχαριστώ θερμά. για την συμμετοχή σας στη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στο σημείο 5, ενδιάμεση αναθεώρηση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Okay, dann würde ich äh, als ersten jetzt der Ας ακούσουμε αν δεν έχετε αντίρρηση τώρα την Επιτροπή πρώτη να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της αναθεώρησης. Κυρία Κιμπέροβα είναι εδώ. Παρακαλώ, εσείς τώρα. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομα θα σας παρουσιάσω το έγγραφο που εξέδωσε η Επιτροπή στις 10 Αυγούστου φέτος. Πρόκειται για την ενδιάμεση αναθεώρηση ε, για το ε, ε, πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη. Πολύ σύντομα να σας πω ότι όπως γνωρίζετε έχει μεγάλη σημασία η έρευνα και η ανάπτυξη για την καινοτομία βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγικής 2020 και ε, στόχος ε, είναι να αντιπροσωπεύει το 3% του ε, ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Επίσης η Ένωση Καινοτομίας είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες για το 2020. Τι ακριβώς λοιπόν είναι το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Θέτει τις ε, προϋποθέσεις που θα πρέπει να σέβονται τα κράτη-μέλη όταν ε, παρέχουν ε, κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Τίθενται λοιπόν οι προποθέσει πλαίσιο για τα κράτη-μέλη για το πώς θα δαπανούν τα χρήματά του για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και θα είναι συμβατό με την κοινή αγορά. Υιοθετήθηκε υπό, ε, το, υιοθετήθηκε στα πλαίσια ε, ενός γενικότερου πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που ξεκίνησε η Κομισιόν το 2005 που στόχο είχε να διοχετεύονται οι κρατικές ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς όπως για παράδειγμα την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία ή το περιβάλλον ε, κλπ. Ένας από τους στόχους της ε, μεταρρύθμιση αυτής ήταν ε, να υπάρχει καλύτερη ε, οικονομική υποστήριξη όσον αφορά τις, τους υπολογισμούς των κρατικών ενισχύσεων. Το πλαίσιο προβλέπει ενδιάμεση αναθεώρηση Ε, και αυτός είναι ο λόγος ε, που δημοσιεύθηκε το έγγραφο αυτό φέτος. Ε, θα πρέπει να το δείτε αυτό κυρίως ω ένα έγγραφο που εξετάζει την κατάσταση και την εφαρμογή του πλαισίου. Δεν πρόκειται για μέρο τη αναθεώρησης, πρόκειται απλά για την κατάσταση των πραγμάτων. Η αναθεώρηση θα ξεκινήσει τώρα το φθινόπωρο ε, βρισκόμαστε λοιπόν δύο χρόνια πριν τη λήξη του, διότι λήγει το 2013 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ξεκινήσει μια ευρία ε, δημόσια διαβούλευση φέτος στο φθινόπωρο με βάση ένα ερωτηματολόγιο που θα δημοσιευθεί. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια σχετικά με την ε, πολιτική για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι οι κρατικές ενισχύσεις αποτελούν μόνο ένα στοιχείο της πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν άλλα μέτρα στήριξη, ε, τα οποία να μην ε, αποτελούν κρατικέ ενισχύσει, ε, για παράδειγμα γενικά μέτρα τα οποία να ισχύουν για όλε τι επιχειρήσει ή μπορούν να υιοθετήσουν άλλε πρωτοβουλίε πολιτική, όπω για παράδειγμα την προώθηση εταιρικών σχέσεων γνώση. Πρόκειται λοιπόν απλά για ένα στοιχείο τη γενικότερη πολιτική για τι κρατικέ ενισχύσει. Οι κρατικέ ενισχύσει είναι συμπατέ με την εσωτερική αγορά εάν στοχεύουν στην αύξηση της ε, έρευνας και της ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούν ε, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που να αντίκεινται στο κοινό όφελος. Ε, πρόκειται λοιπόν για εξισορρόπηση των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων το πλαίσιο. Αυτό υιοθετήθηκε το 2006 και αύξησε τις ανάγκες των δυνατοτήτων των κρατών μελών ε, να παρέχουν κρατικέ ενισχύσεις ε, για την ε, έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και εισήγαγε την έννοια αυτή της ενίσχυσης για την καινοτομία. Οι υπολογισμοί τώρα ε, γίνονται με τρόπο που να αποφεύγεται το στρεβλωτικό αποτέλεσμα. Προβλέπεται λοιπόν τώρα πια, προβλέπονται δύο είδη υπολογισμών. καταρχήν γίνεται ο υπολογισμός σε σχέση με τα ε, κανονικά μέτρα και επίσης μια, προβλέπεται μια πιο αναλυτική εξέταση των κινδύνων ε, για στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι μέσες κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία αυξήθηκαν ε, μετά την θέση σε ισχύ του πλαισίου αυτού το 2007. Και επίσης, έγινε απλοποίηση ε, του τρόπου που παρέχονται οι κρατικές ενισχύσεων ε, που ε, έγινε το 2008, διότι μεγάλο μέρος των μέτρων που είχαν συμπεριληφθεί στο πλαίσιο συμπεριλήφθηκαν στον νέο σχετικό κανονισμό και γι' αυτό τα μέτρα αυτά που συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό GBR επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρο των επενδύσεών του ε, στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία χωρί ε, κοινοποίηση προ την Κομισιόν. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικό βήμα απλοποίηση τη διαδικασία ε, για τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια τώρα σχετικά με τις εμπειρίες μας Ουσιαστικά είδαμε ότι το παρόν πλαίσιο μέχρι τώρα έχει αποτελέσει χρήσιμο ε, ε, εργαλείο για ε, πιο καλά στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον αριθμό των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν εντός του πλαισίου και του σχετικού κανονισμού. Τα κράτη-μέλη τώρα πια έχουν αρκετέ εμπειρίε ε, με την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Η νέα αυτή αναλωτική ε, ε, ο νέος αυτός υπολογισμός φαίνεται να έχει θετικές επιπτώσεις και εξασφαλίζει οι κρατικές ενισχύσεις ε, να αποτελούν κίνητρο για τις επιχειρήσεις. Επίσης, οι κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται μέσω του πακέτου αυτού ε, είναι αρκετά χαμηλές σε σχέση με τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν από όλα αυτά. Θα ήθελα να σας ε, πω λίγα λόγια για την ε, αναθεώρηση ε, του πλαισίου αυτού που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Καταρχήν λοιπόν θα πρέπει να επιδιώξουμε ε, ε, διασαφήνιση και ερμηνεία των ε, κανόνων, διότι λαμβάνουμε αρκετά σχετικά ερωτήματα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Θα το εξετάσουμε αυτό περαιτέρω. Επίσης θα πρέπει να εξεταστούν νέοι πιθανοί τομείς για παράδειγμα, θα πρέπει να εξεταστούν ε, οι key enabling technologies, οι ε, βασικές τεχνολογίες ε, γενικής εφαρμογής. Ε, ξέρω ότι υπάρχει, ε, ότι εκπονείται σχετική έκθεση, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα συμπεριλάβουμε τα αποτελέσματα της στην αναθεώρησή μας. Επίσης φαίνεται ότι οι δυνατότητες που προσφέρει το πλαίσιο και ο σχετικός κανονισμός, κανονισμός δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη-μέλη. Ε, οι κρατικές ενισχύσει, δηλαδή παραμένουν ε, κάτω, του ε, κάτω από το ανώτατο όριο. Θα το εξετάσουμε και αυτό λοιπόν στα πλαίσια της ανθεώρησης. Επίσης εξετάζεται και το θέμα των αυπηγείων, διότι το σχετικό πλαίσιο περιέχει ε, ένα σχετικό στοιχείο και θα αναθεωρηθεί επίσης. Το κομμάτι της καινοτομία λοιπόν που αφορά τα ναυπηγεία θα μπορούσε να, χρησιμοποιηθεί, να ενταχθεί στο πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη επίσης. Όπως σας είπα η αναθεώρηση θα ξεκινήσει τον, το φθινόπωρο. Η Κομισιόν πολύ ευχαρίστω θα σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με τα μελλοντικά βήματα στη διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή τη και επί τη ευκαιρία τη παρουσίας σα, θα εντυπώσω κάποιες ερωτήσεις σε εσά για κάποια από τα ζητήματα του κειμένου αξιολόγησης. Πρώτη ερώτηση. Στο έγγραφο της Επιτροπής λέγεται ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα σχετικά με το, τους τομείς της έρευνας, ε, της καινοτομία και της έρευνας και θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ενώ άλλες επενδύσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ε, τον τρόπο να αλλάξει αυτό το σύστημα. Λέτε λοιπόν ότι, λέει η Επιτροπή, το 2010-2011 το 90% των κρατικών επιχορηγήσεων απορροφήθηκε από τις μικρές επιχειρήσεις. από τις μεγάλες επιχειρήσεις και ότι δεν έχουν ε, αρκετό, ε, αρκετή παρουσία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες όμως αποτελούν την ε, σπονδυλική στήλη, τη ραχοκοκαλιά της ε, οικονομίας μας και ασφαλώς θα πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο σε, αυτή, την, σε αυτές τις ενισχύσεις. Αφού λοιπόν Έχουμε αυτά τα δεδομένα. Δεν θεωρείτε ότι είναι υπερβολικός ο γραφειοκρατικός φόρτος για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε ε, επιλογές οι οποίες θα βοηθούσαν περισσότερο τις μικροπιστές επιχειρήσεις, θα ελάφρυναν αυτόν τον γραφειοκρατικό φόρτο. Παρακαλώ η Επιτροπή για να απαντήσει. Ναι, αυτό που είπα για την ερώτηση σου Όπως είπα λοιπόν θα γίνει η σχετική προσαρμογή και η συζήτηση για την ερμηνεία συγκεκριμένων άρθρων, αλλά πάντως είναι πολύ σημαντική η δημόσια διαβούλευση στο άδειο αυτό για μας, γιατί βλέπουμε και πολύ σημαντικέ ε, επεμβάσει από τα κράτη-μέλη, από τους εμπλεκόμενου. στον κλάδο. Και άρα δεν μπορούμε να έχουμε απαγειωμένες θέσεις αυτή τη στιγμή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούμε βέβαια να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες με λεπτομέρειες και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα ακόμα να συμπληρώσω ότι το πλαίσιο στο οποίο αναφέρομαι ορίζει κάποιες συνθήκες που ε, μπορούν να αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Το πώς θα τις αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη είναι δική τους ε, ευθύνη το πώς θα δαπανίσουν τους, τα χρήματα για να επιτύχουν τους στόχους, δηλαδή ή ποιους στόχους θα ε, εξυπηρετήσουν κατά προτεραιότητα. Και βέβαια κάποια από εσά σε μεγάλο βαθμό ε, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ω κρατικέ επιδοτήσει. Εν πάση περιπτώσει όμω είναι ζήτημα των κρατών μελών το πώ θα αξιοποιήσουν τα κονδύλια αυτά. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Ρόιλ, για τι απαντήσει σα. Δεν βλέπω να ζητεί κανεί άλλο το λόγο. Και άρα μπορούμε να κλείσουμε και αυτό το σημείο τη μισή διάταξη. Στο επόμενο δεν έχω τίποτε στα διάφορα. Προσεχή συνεδρίαση 19 Σεπτεμβρίου. Και με χαρά θα σας ξαναδώ και πάλι. Ευχαριστώ και χαίρετε.